Ladies and gentlemen, may I ask you to take your... Καθίστε παρακαλώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως. I open the regular meeting of Regi Committee. Κηρύττω λοιπόν την έναρξη της συνεδρίασης. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημέρησης διάταξης. Μπορούμε να τη δεχτούμε όπως είναι όπως έχει. Δεν έχετε σχόλια, δεν έχετε παρατηρήσεις, αντιρρήσεις. Ευχαριστούμε. Εγκρίνεται. Έγκριση των πρακτικών της ε, 17 Σεπτεμβρίου 2015 είναι διαθέσιμα επιγραμμικά γιατί όπως θυμάστε αποφασίσαμε να, να είμαστε λίγο πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και να μειώσουμε την εκτύπωση εγγράφων. Όπως πάντα λοιπόν, αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θα θεωρηθούν τα πρακτικά ότι έχουν εγκριθεί. Τρίτο σημείο είναι οι ανακοινώσει της Προέδρου. Από, καταρχήν από τη συνεδρίαση των ε, επικεφαλής των Επιτροπών με το Σώμα των Επιτρόπων που έλαβε χώρα στο Στασβούρο σε 7 Οκτωβρίου. Η συνέλευση των Πρόεδρων των Επιτροπών έκανε την ετήσια της ε, συνάντηση με τους Επιτρόπους για να εξεταστεί το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για του χρόνου. Ήταν και νέο το σχήμα αυτής της ε, συνάντησης. Αντί να είναι παρόντες και οι συμπρόεδροι, έγιναν οι συζητήσεις σε συμπλέγματα, σε ομάδες επιτροπών που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα και μόνο το βράδυ έγινε μια συνεδρία σε ολομέλειας με όλες τις επιτροπές παρούσες. Εγώ ήμουν στο σύμπλεγμα Α, Εργασίας, Ανάπτυξη και Επενδύσεις, που περιλάμβανε 10 επιτρόπους και 8 επικεφαλής επιτροπών. Στην Πρόεδρευση ο κύριος Αρτουή από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και τον ε, Αντιπρόεδρο Κατάινεν της Κομισιόν. Εγώ έλαβα το λόγο σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής συνοχής. Η Επίτροπος Γεωργίευα ανέφερε ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση της Κομισιόν το 2016 που θα εστιάζει στην προσαρμογή του πολιετούς πλαισίου με τις προτεραιότητες σε επίπεδο πολιτικής. Θα δοθεί έμφαση στην απόδοση, στην απλοποίηση, επίσης που είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Σικέρσκι από την Επιτροπή Γεωργίας <clears throat> και μεγαλύτερη λογοδοσία. Στην Ολομέλεια υπήρξαν εκθέσεις από κάθε σύμπλεγμα από την κυρία Γκρέσλε, την πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, που ήταν συνεισήγητρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σύμπλεγμα Α. Ο κ. Κατάινεν τόνισε ότι είναι σημαντική η διοικητική απλοποίηση για όλα τα ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμά μας λοιπόν για την απλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλειών έγινε ακουστό στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη παρατήρηση, η πρώτη ανακοίνωση που ήθελα να σας κάνω. Δεύτερον υπήρξε μια άτυπη Υπουργική Σύνοδος υπό την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Προβλέπεται να εξεταστεί στη συνάντηση των συντονιστών. Μετά από την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ζηρά στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας μπορώ να σας πληροφορήσω για την άτυπη αυτή Υπουργική Σύνοδο που θα κάνει η <clears throat> Προεδρία του Λουξεμβούργου. 13 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αντιμετώπισε την πολιτική συνοχής εδώ όμως δεν υπήρχε παρουσία εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ήμασταν προσκεκλημένοι. Θα γίνει λοιπόν αυτή η άτυπη συνεδρίαση υπουργών στις 26 Νοεμβρίου για την χωροταξική σχεδίαση και, και επίσης 27 Νοεμβρίου. Και εγώ έχω προσκληθεί για να λάβω το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής μας και έχω δεχτεί αυτή την πρόταση, οπότε θα υπάρξει εκπροσώπησή σας κατά τη διάρκεια της άτυπης Υπουργική Συνόδου στο Λουξεμβούργο. Τρίτη, τρίτη ανακοίνωση για τη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου ήμουνα μαζί με τον κύριο Κατάινεν συμπρόεδρη. Έγινε αυτό στα πλαίσια της, ε, των ανοιχτών ημερών της Επιτροπής των Περιφερειών με συμμετοχή της Επιτροπής μας. Τα κύρια θέματα ήταν η εφαρμογή των αρχών εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τι εταιρικέ σχέσει και τα λειτουργικά προγράμματα, απλοποίηση τη εφαρμογή τη πολιτική συνοχή, η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στην πολιτική συνοχή Συνέργειας μεταξύ των διαφόρων εργαλείων και των ταμείων για στρατηγικές επενδύσεις και αναφέρθηκε επίσης μια σχεδιαζόμενη κοινή δήλωση των δύο επιτροπών σε σχέση με, την, με το θεματολόγιο του αστικού χώρου. Συζητήθηκε στη συνέχεια το θέμα αυτό, θα συζητηθεί μάλλον και θα γίνει μια πρόταση προς εσάς από τους συντονιστές. Τελευταίο αλλά όχι ίστατο σημείο Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Όμερζε να μας κάνει μια σύντομη ενημέρωση για την αποστολή μας στην Σικελία. Έχετε το λόγο κύριε Όμερζε. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα με κατηγορήσω να ενημερώσω την Επιτροπή μας σχετικά με τα αποτελέσματα της αποστολής ε, που κάναμε στην Σικελία προέβω μερικών εβδομάδων. Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από το σύνολο των μελών των πολιτικών ομάδων και εγώ ήμουν επικεφαλής, είχα αυτή την τιμή και πήγαμε στην Κατάνια Πέραν των ε, θεμάτων που μας απασχόλησαν, πήγαμε στην ε, Σικελία και αντιμετωπίσαμε το καυτό πρόβλημα της επικαιρότητα, δηλαδή η κρίση των ε, προσφύγων. Και διαπιστώσαμε σε ποιο σημείο οι αρχές της Σικελίας καταβάλουν και κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να ε, αντιμετωπίσουν σύμφωνα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο και να μπορούν έτσι να υποδεχθούν τους ε, μετανάστες. Το συζητήσαμε λοιπόν ε, το ζήτημα και είδαμε επίση τις δυνατότητες που μπορούν να υφίστανται στο πλαίσιο του κανονισμού περί συνοχής ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις περιφέρειες ε, που πρωτίστως αντιμετωπίζουν αυτήν την ροή των μεταναστευτών, μεταναστών. Συζητήσαμε με τον ε, αρμόδιο υφυπουργό της Ιταλίας, ε, τον οποίο, τον συζητήσαμε στο πλαίσιο μιας βίντεο διάσκεψης, και μας ανέφερε για τις εργασίες που έχουν αναλάβει αλλά και εμείς συζητήσαμε για το θέμα αυτό και ειδικά για μια ρήτρα περί μετανάστευσης που θα στηρίξει αυτές τις προσπάθειες και ταυτόχρονα να απαλλάξει τα κράτη που καταβάλουν προσπάθειες από μια σειρά κανόνων σε θέματα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Όλα αυτά λοιπόν πάντω βρίσκονται ακόμα επιτάπητο. Τώρα, για να επανέλθουμε στο Σικελία, αντικείμενο τη επισκεψή μα ήταν να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διαφορετικών Ταμείων για το 2020 και για να λάβουμε υπόψη την περίοδο 2007-2013 και να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τις σικελικές αρχές για τις ε, εξελίξεις και τις δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω δύο πράγματα. Τα χαρακτηριστικά της Σικελίας, μια νησιωτική περιοχή, μια περιοχή που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες ε, στην Ευρώπη, καθιστά ιδιαίτερα περίπλοκο, αυτή τουλάχιστον είναι προσωπική άποψη, την εφαρμογή των νέων στόχων που έχουν τεθεί με Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς πρέπει να καταβληθούν λοιπόν, περαιτέρω προσπάθειες για να καλύψουν τις καθυστερήσεις και είναι γεγονός ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν ακόμα υπάρχει ανάγκη για πολλές ε, επενδύσεις στις υποδομές. Η Σικελία όπως και άλλα ε, και νησιωτικές περιοχές έχουν ανάγκη να ξεπεράσουν αυτήν την ε, νησιωτικό χαρακτήρα τους και αυτή είναι, είναι μερικές από που κάναμε που σήμερα έχουμε και τα θέματα της καινοτομίας όπου διαπιστώσαμε πως σε ζητήματα έρευνας, καινοτομίας, σύνδεσμους και σχέσεις με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν αναλυφθεί μεγάλες προσπάθειες, θεωρώ ότι βρίσκονται στον σωστό δρόμο και οι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί μια ε, ενοποιημένη νησιωτική πολιτική. Ευχαριστώ λοιπόν το σύνολο τη ε, υπηρεσία μας ε, και του προσωπικού μα που φρόντισε να πραγματοποιηθεί σε πολύ καλό κλίμα και κατά από τις βέλτιστες δυνατότητες που υπήρξαν για την διεξαγωγή αυτής της Ευχαριστώ πολύ. Έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το ε, σημείο 3 της Μέσης Διατάξεως, ανακοινώσει του Προέδρου και να συνεχίσουμε την Μέση Διάταξη. Επόμενο σημείο Αυτή είναι η Συμφωνία στρατηγική σχέση για την Πολιτική Συνοχή. Σήμερα έχουμε την ε, ευκαιρία να ακούσουμε μια παρουσίαση εξωτικής μελέτης θέμα επανεξέταση των συγκεκριμένων συμφωνίων εταιρική σχέση. Η Επιτροπή μα αποφάσισε πέρυσι να ζητήσει μια ε, ε, έκθεση για το ζήτημα αυτό μετά από προκήρυξη διαγωνισμού και ζητήσαμε από την ε, εταιρεία ΜΕΤΙΣ να αναλάβει αυτήν την μελέτη. Όπου περιλαμβάνεται μια συνεκτική ανάλυση της, του θέματος των συμφωνητρικής σχέσεων, το Κοινοβούλιο κατά διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το, και το νομοθετικό πλαίσιο. Και αναφέρεται στους ε, θέμα των συμφωνιών και της ε, σύμπτωσης με τη Ζωτική 2020. Ανάμεσά μας βρίσκεται η κυρία Ιζαμπέλ Νέιλαν, από την επιτερία Μέτης που θα παρουσιάσει την μελέτη και μια που θα το συνδυάσουμε με την παρουσίαση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειών επί του αυτού θέματος. Θα τη ζητήσω λοιπόν να λάβει το λόγο για ε, το πολύ 10 λεπτά αν είναι δυνατόν και μετά θα ακούσουμε την Επιτροπή των Περιφερειών και θα περάσουμε στην, ε, στο γύρο των ερωταποκρίσεων. Κύριε Νέιλον, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τη μελέτη. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο στι διαπραγματεύσει για, για τη σύναψη των εταιρικών σχέσεων, που είναι η συμφωνία ουσιαστικά μεταξύ τη Κομισιόν και των κρατών μελών για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και, των, και του Ταμείου Επενδύσεων για να υπάρξει ε, φυγράμιση των, ε, της χρήσης των ταμείων με τους ε, στόχους 2020 και τους στόχους βεβαίως που απορρέουν από τη συνθήκη. Η μελέτη αυτή λοιπόν πραγματεύεται αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Αυτό που θα κάνω σε αυτή την παρουσίαση και θα προσπαθήσω να μείνω εντός των 10 λεπτών είναι να σας παρουσιάσω συνοπτικά το περιεχόμενο και τους στόχους των, της μελέτης, να σας δώσω μια πρώτη γεύση μετά θα σας μιλήσω ε, σύντομα για τα μεθοδολογικά σημεία, τα βασικά θέματα στα οποία, με τα οποία ασχολήθηκε η μελέτη και μετά θα μπούμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες για κάποια από αυτά τα σημεία τα οποία ε, ήταν σημαντικά για το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ο στόχος λοιπόν όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, ήταν να παρουσιάσουμε μια συνοπτική και συνθετική ανάλυση της, ε, των υιοθετηθήσεων ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης. Εδώ έχουμε δηλαδή και μια γενική εικόνα όλων των ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης που υπάρχουν προς το παρόν και ο στόχος είναι να τονίσουμε από τη μία το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων και να δούμε και τη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις, τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές διατάξεις. Επίσης, παρέχουμε μια σύντομη γενική εικόνα των στρατηγικών επιλογών πολιτικής που, που κάνουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια αυτών των εταιρικών σχέσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Και επίσης δίνεται και κάποια έμφαση σε όσα αφορούν στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, μέθοδο τη διερευνητική που ε, ε, κάναμε, ήταν έρευνα που έγινε σε επίπεδο κρατών μελών, από, τις, από τα γραφεία των κρατών μελών. Κάναμε λοιπόν συντηρητική ανάλυση των 28 PAs και βεβαίως χρησιμοποίησαμε και άλλα επιλεγμένα έγγραφα, είδαμε τα CSR, τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τα εθνικά στρατηγικά έγγραφα, τα έγγραφα θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις εταιρικές σχέσεις και στη μελέτη έχουμε ολοκληρωμένες ε, ε, περιλήψεις ε, και βεβαίως υπάρχει και η πιο λεπτομερής εκδοχή αυτών στο παράρτημα. Οι εταιρικές σχέσεις, οι συμφωνίες εταιρικές σχέσεις είναι βεβαίως στη γλώσσα του κράτους μέλους και φυσικά η πρόκληση ήταν να μελετήσουμε όλα αυτά τα κείμενα στις διάφορες γλώσσες που είναι γραμμένα χρησιμοποιώντας βεβαίως ε, ένα μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων για να το κάνουμε αυτό και μετά να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις επιμέρους ε, εκθέσεις για να καταλήξουμε σε μια οριζόντια και πλήρη ε, ανάλυση όλων αυτών των PAs. Βεβαίω δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ομοιογένεια στο πώ περιγράφουν τα έγγραφα αυτά των πρωτομελών τα στοιχεία κλειδιά στα οποία περνάω τώρα και βεβαίω ο κατάλογος που σας αναφέρω δεν είναι διεξοδικό, γιατί οι εταιρικέ σχέσεις καλύπτουν πολύ περισσότερα σημεία από αυτά, αλλά αυτά ζητήθηκε να μελετήσουμε. Καλύψαμε λοιπόν ουσιαστικά το, ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα, την θεματική συγκέντρωση, είδαμε την αφιγράμμιση των PA και, των, ε, και της 2020, είδαμε τη διαφάνεια της διαδικασίας, τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη ενσωματώνουν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης αυτές τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, μελετήσαμε τις συνέργειες μεταξύ της χρήσης των ε, Διευθυντικών Ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης. Είδαμε συνολικά τα εξάντε αιρεσιμότητα και πώς αυτή παρουσιάζεται στα πλαίσια των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και επίσης είδαμε και κάποιες συγκεκριμένε διατάξεις που έχουν να κάνουν με δημογραφικές προκλήσεις και απλούστευση αλλά και ηλεκτρονική συνοχή. Τώρα, για το, για το γενικό πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη θεματική συγκέντρωση. Και τα 28 κράτη-μέλη έχουν, ε, χρησιμοποιούν τα τρία ταμεία, το ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνική Συνοχή ε, και το Ανάπτυξη Πέθρου. Ε, οι 20 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα, τα πολυταμιακά επιχειρησιακά προγράμματα σε αυτή την προγραμματική περίοδο συνδυάζοντας βεβαίως ε, τα, ταμεία από τα, τα κονδύλια από τα διάφορα ταμεία, άλλοι συνδυάζουν το ERDF με το Ταμείο Συνοχής, 11 ε, κρατημέλη, 7 ε, κρατημέλη κρατούν, συνδυάζουν και τα τρία ταμεία και υπάρχουν 8 κρατημέλη τα οποία έχουν μονοταμιακά προγράμματα. Αυτό έχει να κάνει με το σύστημά τους, γιατί δεν, ε, δεν έχουν τόσο τομεακή ας πούμε, προσέγγιση. Και είναι και αρκετά έτσι, σκεπτικοί σε ό,τι αφορά το, τη χρήση του μονοταμιακού προγράμματος, γιατί θεωρούν ότι η χρήση πολυταμιακού προγράμματος μπορεί να είναι πιο ε, γραφειοκρατική. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα επίσης θεματικής συγκέντρωσης. Το Ταμείο Ανάπτυξη Πέθρου αφορά ε, στους πρώτους τέσσερις στόχους. Υπάρχουν 11 συνολικά. Οι πρώτοι τέσσερις είναι αυτοί στους οποίους ε, ε, επικεντρώνεται το ταμείο αυτό, το RTDI, το ICT, οι μικρομεσαίες και το διεξόδιο του άνθρακα. Το κοινωνικό ταμείο ασχολείται με τους στόχους 8, 9, 10 και 11, απασχόληση, φτώχεια, διαβίου μάθηση και διοικητικές δυνατότητες. Και αυτό που, ε, και επίσης υπάρχουν και ε, κάποιοι κανόνες. 20% ας πούμε της ε, χρηματοδότησης πηγαίνει στον στόχο 9 για τη φτώχεια και 5% στην βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω αυτών των δομών λοιπόν τα κράτη-μέλη διάλεξαν τους θεματικού τους στόχους και μάλιστα 28, και τα 25 μάλλον επέλεξαν και τους 11 στόχους και, και μόνο τρία επέλεξαν κάποιους από αυτούς. Εδώ σας δείχνω μια γραφική παράσταση για να δείτε συνολικά τη χρήση των ταμείων ανάλογα με θεματικό στόχο. Όπως βλέπετε, ε, ο 6, ο 7 και ο 3 είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ε, οι μεταφορές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, η εξάντε ερεσιμότητα. Όλα τα κρατημέλη πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες ε, περιγράφουν στα, ε, στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, με διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας στο καθένα. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι οι περισσότερες, ε, και οι γενικές δηλαδή, και οι ε, τομεακές προϋποθέσεις πληρούνται στην, στα 15, στην Ευρώπη των 15, και τα νεότερα κρατημέλη, όσο νεότερα είναι τα κρατημέλη, τόσο λιγότερες είναι οι προϋποθέσεις που πληρούνται. Σε ό,τι αφορά τώρα τους στόχους, τα θέματα μάλλον, το υψηλότερο επίπεδο πλήρωσης είναι η προσαρμογή στην ε, μενομοθεσία για το περιβάλλον και το χαμηλότερο είναι στα ε, στατιστικά συστήματα. Αυτό βέβαια εξηγείται γιατί τα κράτη-μέλη ε, ευθυγραμμίζουν τα, τα συστήματα τους αυτά, τα στατιστικά, με το σύστημα της Κομισιόν. Οπότε τα προσαρμόζουν όσο προχωρούν και όσο πιο επιχειρησιακά γίνονται τα συστήματα, όσο προχωρούν τα προγράμματα, τόσο περισσότερο και τα συστήματα πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Όλα τα κράτη-μέλη περιμένουν ότι θα, πληρούν, θα πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις πριν την ε, προθεσμία, που είναι ο Δεκέμβριος του 2016. Επίσης, παρουσιάσαμε το επίπεδο αυτό, τις ε, επιτυχίες αυτού, αυτής στο γραφικό αυτό σχήμα που βλέπετε. Κάποιοι, έχουν, ε, ε, κάποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις, κάποιοι όχι. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Και σε ό,τι αφορά τα θεματικά, τις θεματικές ενότητες, βλέπετε πάλι πώς πληρούνται ή όχι ή μερικώς οι ε, προϋποθέσεις αυτές εξάντε. Βεβαίω αυτό αλλάζει όσο τα κράτη-μέλη προχωρούν τα προγράμματα και επιτυχάνουν τους στόχους, βεβαίως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να ενημερωθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ηλεκτρονική συνοχή και την απλούστευση, αυτό ήταν ένας από τους βασικούς τομείς, πυλώνες της απλούστευσης, η ηλεκτρονική συνοχή. Ε, το σύστημα αυτό υπήρχε και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και τα κράτη-μέλη απλώς τα εξελίσσουν περαιτέρω, τα ευθυγραμμίζουν περαιτέρω για να ευθυγραμμιστούν με το SFC, το πρόγραμμα της Κομισιόν για τούτη την προγραμματική περίοδο. Οι συμφωνίε Εστερικής Σχέσης περιγράφουν πολλές φορές με πολλές λεπτομέρειες άλλες με λιγότερες ε, τα τεχνικά στοιχεία αυτού του συστήματος και αυτό που περιλαμβάνει ή τέλο πάντων αυτό που θεωρούμε ότι είναι η, η ηλεκτρονική συνοχή, είναι οι δικαιούχοι να υποβάλουν τι προτάσει του και τι αιτήσει του μέσω ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένε ιστοσελίδε για του δικαιούχου ε, και του τούντε και υπάρχουν και κάποια κεντρικά συστήματα πληροφορική. Κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν και, πληρο... και περιφερειακά συστήματα. Λοιπόν, μάλλον τελειώνει ο χρόνο μου, οπότε πρέπει να τα πω πολύ γρήγορα τα τελευταία που θέλω να πω για τις συγκεκριμένες ε, ε, προσεγγίσεις, το CLLD και το ITI. Ε, έχουν περιγραφεί παντού ε, τα CLLDs είναι η ε, τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και υπάρχει και στα 28 κράτη-μέλη από τα πολυταμιακά προγράμματα. Στις περιγραφές των κρατών μελών αυτές οι δράσεις χρησιμοποιούνται για να ε, χρηματοδοτηθούν τοπικές ομάδες δράσης στα πλαίσια και της περιφερειακής ανάπτυξης. Και ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση ε, περιγράφεται σε 20 κρατη στα επιχειρησιακά του προγράμματα και καλύπτει κυρίως ε, την ε, αστική πτυχή και βεβαίως καλύπτεται πάλι από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Φτάνω στην τελευταία διαφάνεια, εταιρικές σχέσεις και συντονισμός, όπως περιγράφεται και στη Συμφωνία Εταιρικές Σχέσεις. Αυτή η οριζόντια αρχή έχει υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη και οι συμφωνίες αυτές ε, παρέχουν πληροφορίε, ε, ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετέχουν, ποια είναι τα συντονιζόμενα υπουργεία. Υπάρχει λοιπόν πλήρης περιγραφή σε όλες τις συμφωνίες τερικής σχέση. και βεβαίω αυτό αποτέλεσε τη βάση της δικής μας μελέτης. Επίσης, η δημόσια διαβούλευση για τι για τις συμφωνίες εταιρική σχέσης επίσης ε, περιγράφεται στα επιχειρησιακά προγράμματα. Κάποια κράτη-μέλη ε, έκαναν περισσότερο διαβούλευση σε επιχειρησιακά προγράμματα και κάποια άλλα όχι. Αυτά από μένα. Σα ευχαριστώ πολύ, Λέκη προέδρο. Ήσασταν πολύ κοντά στο όριο που σας έδωσα, γι' αυτό Ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ φορτωμένη μέρη σε διάταξη και γι' αυτό μετράω και τα λεπτά. Και τώρα έχω τη χαρά να μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Ζάγκα, ο οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία και αυτή έχει εγκρίνει μια γρομοδότηση για το αποτέλεσμα και τα πορίσματα των ε, εταιρικών, των προγραμμάτων εταιρικών σχέσεων. Ο κ. Ζέγκερ ήταν ο εισηγητή για το θέμα αυτό στην Επιτροπή των Περιφερειών και έχω τη χαρά τώρα να του δώσω το λόγο. Για 10 λεπτά και εσεί 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε για να παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σε σχέση με τις συμφωνίες συμμετοχής σε λειτουργικά προγράμματα. Η Επιτροπή ΚΟΤΕΡ, που είναι η Επιτροπή Εδαφικής Συνοχής και ασχολείται με τα θέματα αυτά στην Επιτροπή των Περιφερειών, συνεργάζεται με την Επιτροπή σας πολύ καλά. Ο στόχος αυτής της γνωμοδότησης ήταν να αξιολογήσουμε τις συμφωνίες σύνδεση και τα λειτουργικά προγράμματα από πολλαπλέ απόψει. Από την πλευρά των δικαιούχων για αυτά τα εργαλεία και από την έποψη του τοπικού επίπεδου που είναι αυτό το οποίο φυσικά πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα προγράμματα. Και φυσικά οι τοπικές αρχές είναι αυτές που γνωρίζουν καλύτερα την επιτόπια κατάσταση. Οι συνάδελφοι λοιπόν αυτοί, οι δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι των περιφερειών και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν και εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η Επιτροπή των Περιφερειών επιπλέον έχει κάνει μια <clears throat> δημοσκόπηση στην οποία συμμετέσχαν πάνω από 300 φορείς, κυρίως θεσμοί, φορείς ε, όπως το FMF, και η δημοσκόπηση αυτή μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα ε, της Επιτροπής των Περιφερειών. Και Eurocities. Πρόκειται μία, για μία α, έρευνα εκ των κάτω προς τα άνω για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ε, επιτοπίως και πώς εφαρμόζονται οι συμφωνίες σύνδεσης και τα λειτουργικά προγράμματα. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω μερικά σημαντικά στοιχεία τα οποία και αυτά περιλαμβάνονται στην γνωμοδότησή μας. Και μετά μπορώ να σας δώσω και περισσότερα στοιχεία εάν το επιθυμείτε. Ας περάσουμε στο περιεχόμενο. Αναφέρεται ο θεμελιώδης ρόλος της πολιτικής συνοχής σε ό,τι αφορά την επίτευξη της συνοχής σε εδαφικό επίπεδο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις διαφορές ανάπτυξης, τα χάσματα ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό. Αλλά, <clears throat> σε ορισμένε περιπτώσεις, η ανισομέρεια αυτή μεταξύ των περιφερειών, αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Αυτό το είδαμε καθόλου το μήκος και το πλάτος της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που έχουμε περάσει πρόσφατα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό, στο γεγονός ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να δίδει συνέχεια στις βασικές ανάγκες ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας. Και συγχρόνως θα πρέπει <clears throat> να συνάδει με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταρρυθμίσεις της πολιτικής συνοχής, εδώ υπάρχουν διάφορα καινοτόμα στοιχεία. Κάποια από αυτά τα ακούσαμε από τους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν. Αλλά θα ήθελα εδώ να σταθώ περισσότερο στις σχέσεις σύνδεσης. Έχετε εδώ ένα έγγραφο το οποίο εξετάζουν τα κάτι μέρη σε σχέση με το θέμα αυτό, γιατί οι συμφωνίε σύνδεση είναι μία βάση για όλα τα περαιτέρω που γίνονται. Είναι μία προϋπόθεση για να μπορέσει να ευδοκιμήσει η πολιτική συνοχή. Γιατί υπάρχουν αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλα αυτά τα επίπεδα λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουν και να συντονίζονται για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Είναι πολυεπίπεδη λοιπόν η διαχείριση που σέβεται φυσικά και την αρχή της επικουρικότητας και την ανάγκη να λαμβάνουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες οι οποίες εμφανίζονται και οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιηθούν από αυτά τα προγράμματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο εφόσον φυσικά επιθυμούμε η πολιτική συνοχή να αποδώσει καρπούς σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Όλα τα κράτη-μέλη φυσικά έχουν αυτές τις ε, ενώσεις και αυτές τις ε, συμφωνίες συνδέσεων. Είναι πολύ μορφή όμως η πραγματικότητα των κρατών μελών και αυτό φάνηκε και από τις έρευνες που, που έχουμε διαξαγάγει. Πολλές φορές. Η συζήτηση έχει καταδείξει ότι οι σχέσεις σύνδεσης, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα για κάποιες περιφέρειες. Το 75% των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο μας μας ε, ανέφεραν ότι παρά την συμμετοχή, στη συμμετοχή τους εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες ελλείψεις. Τέλος. Δεν πρόκειται μονάχα για τη συμπερίληψη του τοπικού και του περιφερειακού επίπεδου, αλλά και για την πραγματική συμμετοχή τους σε αυτές τις σχέσεις σύνδεσης που είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Και κάτι ακόμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και αυτό φυσικά συνδέεται με την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αναφέρθηκα στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει πλήξει την Ευρώπη πρόσφατα αυτό. Έχει επηρεάσει το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πολλές φορές έχουν έλλειψη επαρκών πόρων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αυξηθεί η χρηματοδότηση, να αυξηθεί και η πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να επιτρέψουμε και στα επίπεδα αυτά να έχουν νέες πηγές χρηματοδότησης για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις πολιτικές αυτές. Πολλές φορές υπάρχει επικάλυψη στα θέματα αυτά και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς αυτό επηρεάζει το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πώς θα εξελιχθούν αυτά και στο μέλλον, είναι απαραίτητο να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να διαμορφωθεί αυτό το πλέγμα εργαλείων στο μέλλον για να είναι πιο επωφελές. Για μας αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει με συνδυασμό των ταμείων, των διαχωριστικών ταμείων και με την ενέργεια, με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αυτά τα ταμεία φυσικά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο ένα μέρος και μετά σε κάποιο άλλο μέρος. Θα πρέπει να έχουν σαφείς στόχους στους οποίους εξυπηρετούν. Όλο αυτό το καιρό λοιπόν μιλάμε για αυτά τα θέματα τα οποία παραμένουν εκκρεμή ως προς την επίλυσή τους. Πρέπει να απλοποιήσουμε παραδείγματος χάρη τις διαδικασίες. Όλο αυτό το διάστημα το, την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού μιλάμε για την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών. Αλλά η πραγματικότητα μας δείχνει ότι όχι μονάχα δεν απλοποιούνται οι διαδικασίες, αλλά κάθε φορά είναι πιο πεπλεγμένες. Γι' αυτό η εκτέλεση των προγραμμάτων γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη. Έχουμε λοιπόν μία μεγάλη πολυπλοκότητα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και πολλές φορές είναι δύσκολο να υπάρξει μια σωστή εστίαση αυτών των ταμείων και μία διασύνδεση μεταξύ τους ακριβώς λόγω των ε, διαδικασιών που είναι βαριές και χρονοβόρες. Αυτή η απλοποίηση λοιπόν είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν αυτές τις δυσκολίες που βλέπουμε κάθε φορά και περισσότερο στην εφαρμογή των πόρων αυτών που έχουμε από τα διαφορετικά ταμεία. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει υπερβολική μεταφορά των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων στι εθνικέ αρχέ. αν υπάρχει μία μορφή επανεθνικοποίηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε προσεκτικά. Φυσικά, <clears throat> εμεί επικροτούμε τη δημιουργία τη ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση. Ελπίζουμε ότι θα στεφτούν υπό επιτυχία οι προσπάθειε τη ομάδα αυτή, ώστε η πολιτική συνοχή τελικά να μπορέσει να αποδώσει τα απαιτούμενα. Χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τις ικανότητες διαχείρισης είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά την διαχείριση των προγραμμάτων αυτών και είναι απαραίτητο να είμαστε σε θέση να δίνουμε την απαραίτητη τεχνική αρρωγή στα κράτη-μέλη. Αλλά είναι πάρα πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Κλείνω πάλι. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και σε ένα ακόμα σημείο. Πρόκειται για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται εκ των προτέρων, εξάντε. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση για την ε, παροχή των απαραίτητων εγγράφων, της απαραίτητης τεκμηρίωσης. Αυτή η καθυστέρηση φυσικά έχει επιπτώσεις και στην εκτέλεση των προγραμμάτων. Σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται στο τρέχον, στο νέο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι μεγάλη καθυστέρηση είναι υποχρεωμένο το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο να αναμένουν για να μπορούν να έχουν την προσθεθέμενη αξία που θα πρέπει να αποκτήσουν από τα προγράμματα αυτά. Επίσης για τις εσωτερικές διαπραγματεύσεις υπάρχει πρόβλημα όταν δεν, το, δεν σέβονται οι αρχικές αρχές τα χρηματοδοτικά πλαίσια. Είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο λόγω της λειτουργίας του εθνικού επίπεδου το περιφερειακό επίπεδο να φύγεται. και επίση σε ό,τι αφορά το σύνολο τη πολιτική συνοχή. Είναι μια πολυεπίπεδη <clears throat> πολιτική, μια διαμεθοριακή πολιτική που χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία CLLD παραγματικά χάρη και είναι επίση μια πολιτική η οποία πρέπει να έχει περιφερειακό χαρακτήρα και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο να είναι. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ορισμένε πολιτικέ οι οποίε ε, αναδύονται και οι οποίε έχουν σαν στόχο να ξαναγίνει συγκεντρωτική διαχείριση αυτών των προγραμμάτων και των πολιτικών. Γιατί με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η σωστή εφαρμογή των εργαλείων περιφερική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα ήρθε η ώρα για να περάσουμε στη ζήτηση. Θα ήθελα να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας σε ένα λεπτό έκαστος. Δεν υπάρχει κάποιος κατάλογος αγορητών, υπάρχει κάποιος εξημών που θέλουν να λάβουν το λόγο. και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εξαιρετική εργασία που κάνατε και ως Επιτροπή των Περιφερειών. Τρία σημεία θα ήθελα να δείξω. εν συντομία. Σε ένα από τα συμπεράσματα της εκθέσεως, κύριε Νίλ, μιλάτε για το διοικητικό άχθος το οποίο θα μειωθεί λόγω της ε, ε, συγκέντρωσης που και να συμβεί σε κάποια κράτη-μέλη. Γιατί λοιπόν αυτό το διοικητικό άχθος θα μειωθεί και περιμένετε αύξηση αυτού του διοικητικού άχθους σε χώρες όπως η Γερμανία που δεν έχουν τέτοια προγράμματα για κάθε κρατήδιο. Μας πείτε λίγα πράγματα σχετικά με τις διαφορές ε, τις ποιοτικέ, διότι έχετε μια πολύ ποσοτική αντιμετώπιση και τέλος μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για τους ε, κλιματικούς στόχους ε, αν βλέπουμε ότι σε περισσότερα από τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούνται διαφορετικά διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σπόλιο για το λόγο. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε αυτά που μας είπε ο πρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών. Η Επιτροπή των Περιφερειών δήλωσε ότι 70% των απαντώντων σε αυτή την έρευνα θεωρούν ότι στην προπαρασκευαστική φάση των ε, ε, προγραμμάτων οι ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών αρχών ελήφθησαν ε, υπόψη εν μέρη ή και μερικέ φορέ καθόλου. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα κατά την άποψή μου, διότι δεν μπορείτε να παραβλέψετε τις τοπικές και περιφερειακέ αρχέ και τις απόψει τους. Και αυτό είναι το ζούτο προβληματικό, διότι δεν ε, αντιμετωπίζεται αυτό τον τρόπο το ζήτημα των ε, ΣΕΣ και θα ήθελα να ρωτήσω εάν δεν υπάρχει κάποια παραβίαση του ενδοσιακού δικαίου. Εάν δεν εφαρμόζεται αυτή η αρχή και θα ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένο αν η Επιτροπή και άλλοι συνάδελφοι απαντήσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την παρουσίαση της μελέτης, ευχαριστώ και για τα όσα μας είπε η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία όντως ε, άσκησε κάποια κριτική και εγώ παρόμοια σχόλια έχω να κάνω. Διαπιστώνω ότι η μελέτη ουσιαστικά είναι ποσοτική, τονίζει τα ποσοτικά, τις ποσοτικές πτυχές και δεν μπαίνει τόσο πολύ στην ποιοτική πτυχή του πράγματος και στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό σε δύο τομείς έχω, έχω ερωτήματα. Καταρχάς η εξάντε ρεσιμότητα, οι προϋποθέσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα για τις αιτίε, γιατί δεν τηρούνται, γιατί δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και τι κάνουν τα κρατημέλη για να το διορθώσουν και να ε, αρθούν στο ύψος των περιστάσεων γιατί δεν μπόρεσα να το δω έτσι λεπτομερώς, γι' αυτό και ρωτώ. Και σε μια παρόμοια κατεύθυνση για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Είναι σημαντικό και στην μελέτη σας φαίνεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά από ό,τι ξέρετε, ξέρουμε και εμείς από τους εμπλεκόμενους φορείς και όσους ε, συμμετέχουν και από την κοινωνία των πολιτών και από τους κοινωνικούς εταίρους, ότι υπάρχουν ε, διαφορετικά είδη εφαρμογή για να το πω ευγενικά και θετικά, και σε ό,τι αφορά τον ορισμό του τι είναι αυτές οι εταιρικέ σχέσεις, αλλά γενικώ υπάρχει στη μελέτη σας μια πολύ θετική εικόνα της ε, εφαρμογής από τα κράτη-μέλη, κάτι που εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, οπότε θα ήθελα να μου πείτε κάτι επ' αυτού. Ευχαριστώ. Κυρία Μπρέσο, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η ερώτησή μου αφορά στην θεματική συγκέντρωση σε επίπεδο περιφερειών διότι είναι ξεκάθαρο πως ε, αν μιλάμε για μεγάλα κράτη όπου υπάρχει περιφερειοποίηση των ταμείων όπου η θεματική επικέντρωση όπως ε, αναφέρθηκε σημαίνει πως όλες οι περιφέρειες χρησιμοποίησαν όλες ή σχεδόν όλα τα θέματα ή απλά όταν γίνεται η άθρηση των, στις επιμέρους χώρες κάθε περιφέρεια έχει επικεντρώσει τη προσοχή της σε τρία ουσιώδη θέματα, διότι είναι πολύ διαφορετικό. Καταλαβαίνετε ότι σε επίπεδο ε, κράτους ε, η συγκέντρωση δεν υπάρχει, αλλά μιλάμε για προγράμματα που είναι περιφερειοποιημένα. Το ε, ζήτημα είναι εάν σε επίπεδο επιμέρους περιφερειών ε, έχουμε εγγυηθεί την θεματική συγκέντρωση ή όχι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντεμάτο. Κύριε Πρόεδρε. Μερικές σύντομες ερωτήσεις δεδομένου του ότι οι συμφωνίες σχέσει σχέσεις ε, πολύ συχνά είναι ψευδείς ε, εντάξει ο όρος είναι δυνατός ε, αλλά πάρτε τον προσεκτικά εάν όμως εφαρμόζονται στα λειτουργικά προγράμματα διαρωτώ με και ερωτώ την Επιτροπή Περιφερειών επειδή είναι αυτοί που ασχολούνται ιδιαίτερα με την με την περιοχή και είναι εάν θα μπορούσαν να προτείνουν καθηγητές γραμμές ε, καλύτερες. Και να ρωτήσω επίσης ε, σχετικά με τους θεματικούς στόχους, θα ήταν καλύτερο να προτείνουμε στις λιγότερο εμπληκμένες περιφέρειες ε, να επικεντρωθούν σε λίγους θεματικούς στόχους και τέλος σχετικά με την τεχνική αρρωγή τι προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, κάποια περιφερειακά αλλά και εθνικά προγράμματα που προβλέπουν βοήθεια στις ε, διοικήσεις. Αλλά αυτού του είδους η αρρωγή φαίνεται πως έχει, δεν έχει φέρει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα ή τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κυρία Νίλον, μπορείτε να απαντήσετε μέσα σε τρία-τέσσερα λεπτά. Είμαι όσο έτοιμο όσο θα είμαι ποτέ, λέει η κυρία Νίλον, σε ό,τι αφορά το διοικητικό άκθο. Αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει κατανοητό και σας λέω και πάλι κάνουμε έρευνα για τις συμφωνίες εταιρικού χαρακτήρα και δεν ήμασταν σε θέση μέσα στη σύντομη αυτή μελέτη να περάσουμε στο περιφερειακό επίπεδο και να δούμε τι γίνεται σε κάθε συγκεκριμένο επίπεδο. Βλέπουμε τις συμφωνίες αυτές ως πλαίσιο. Για το πρώτο ερώτημα λοιπόν που ετέθη για το διοικητικό άχθος. Υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία στην ε, προγραμματική αυτή περίοδο μεταξύ των οποίων και η μείωση του αριθμού των, ε, προγραμμάτων αυτών Αναφέρεται πραγματικά χάρη το περίπτερο της Αυστρίας. Ενώ υπήρχαν στο παρελθόν εννέα περιφερειακά προγράμματα, τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα μονάχα. Βέβαια συνεχίζεται η ανάγκη συνεργασίας των Λέντερ με, μεταξύ τους στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Είναι ένα νέο σύστημα, δεν είναι πια κάτι το οποίο αναπόκειται σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο εθνικό. Αυτό σημαίνει ότι και οι διαδικασία συντονισμού είναι πιο έντονη. Πρέπει να υπάρξει η συν... συντονισμός μεταξύ των περιφερειών αυτών. Επίσης υπάρχουν <clears throat> προγράμματα τα οποία είναι πιο πολλαπλού χαρακτήρα, αυτό σημαίνει περισσότερο συντονισμό. Υποτίθεται με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει καλύτερο ε, συντονισμό των προγραμμάτων, αλλά αυτό φυσικά απαιτεί περισσότερε συζητήσει, περισσότερε διαπραγματεύσει. Είναι ένα ένας νέος χώρος που είναι ανεξερεύνητος ακόμα για τις ε, εμπλεκόμενες αρχές και για την ποιότητα των συμφωνιών εταιρική σχέση αυτό δεν τολμούμε να το αντιμετωπίσουμε φυσικά. Αλλά η μελέτη μας εστιάζει στο τι έχουν κάνει οι συμφωνίες αυτές μέχρι τώρα, προσπαθήσαμε να δούμε, να δείξουμε τι περιέχουν αυτές οι συμφωνίες, αλλά χρησιμοποίησαμε τις απόψεις πολλών εμπειρογνωμόνων που είχαν διαφορετικές βέβαια θέσεις. Δεν έχουμε καταλήξει σε μια αξιολόγηση των ε, συμφωνιών εταιρική σχέσης. Απλώς το περιεχόμενό τους εξετάσαμε. Δεν θα τολμούσα λοιπόν να προχωρήσω σε μια αξιολόγηση αυτών των συμφωνιών. Κάποια από τα στοιχεία της μελέτης μας δεν ήταν εκτενή ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη η ηλεκτρονική συνοχή κτλ. Δεν είχαμε ε, επεκταθεί σε μεγάλο ε, βαθμό για τα θέματα αυτά. Και γι' αυτό φυσικά δεν τα κράτη-μέλη, ήταν η δομή της ερευνάς μας σε ό,τι αφορά τους θεματικούς στόχους. Σύμφωνο με τον άλλο συνάδελφο που είπε ότι σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο εθνικό, μπορούν να καλύπτονται όλοι οι θεματικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο και παρόλα αυτά να υπάρχει συγκέντρωση σε επίπεδο περιφερειών ιδίως στις χώρες που έχουν πολλά α, προγράμματα αυτού του είδους όπως είναι η Ισπανία <clears throat> αλλά με πολλές περιφέρειες αλλά και οι χώρες με τα λίγα λειτουργικά προγράμματα ή που έχουν λειτουργικό πρόγραμμα, ένα λειτουργικό πρόγραμμα <clears throat> αναταμείο μπορούν να χρησιμοποιούν όλους τους θεματικούς λόγους ε, στόχους μάλλον, <clears throat> ενώ συγχρόνως σέβονται την αρχή της συγκέντρωσης των πόρων όπως απαιτούν οι κανονισμοί. Για την μη τήρηση της εκ των προτέρων ερεσιμότητος, της εξάντερας ερεσιμότητος, ούτε και αυτό ήταν από τα σημεία εστίασης της ε, έκθεσής μας. Γιατί δεν τηρείται αυτή η ερεσιμότητα. Απλώς να δούμε αν τηρείται ή όχι. Έχει γίνει από την DG Regi μια λεπτομερής μελέτη για αυτά τα θέματα και εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά για τις περιπτώσεις που τηρήθηκε το λιγότερο για τα υδάτινα θέματα, για τα απορρίμματα και για τις μεταφορές, εκεί δεν έγινε αυτό δυνατό γιατί δεν υπήρχε ένα γενικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, ή μια πολιτική για τιμολόγηση του νερού ή ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές. Αυτά είναι παραδείγματα για τους λόγους για τους οποίους η εξάντια αιρεσιμότητα δεν μπόρεσε να τηρηθεί. Και εν γέννη για την εξάντια αιρεσιμότητα στα συστήματα πληροφορικής. Αυτά ίσως έχουν επιτευχθεί, έχουν τηρηθεί κανόνες μέχρι τώρα. Αλλά τότε υπήρχαν κάτι κάποια κρατημέλη τα οποία ακόμα ήταν στη φάση της εγκατάστασης των συστημάτων και δεν ήταν έτοιμα τα συστήματα αυτά, απλώς όμως θα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις έτοιμα όταν εφαρμοστούν τα λειτουργικά προγράμματα. Και για την αρχή της εταιρική σχέσης, αυτό το οποίο παρουσιάζουμε εδώ, είναι αυτό το οποίο περιέχονται στις συμφωνίες αυτές καθεαυτές και όχι στην εφαρμογή του. Εμείς, ε, ε, εγώ προσωπικά ασχολήθηκα μόνο με την περίπτωση της Αυστρίας, όπου υπήρχε μεγάλη παρουσία των περιφερειών και σε τοπικό επίπεδο υπήρχε παρουσία και ένα μεγάλο φάσμα ε, κοινωνικών εταίρων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μάλλον μη, κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ατόμων με αναπηρίες κτλ, τμήματων της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν τα μελετήσαμε, σε ό,τι αφορά την διατύπωση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία να σας δώσω σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμοστήκαν όλα αυτά στην πράξη. Νομίζω ότι καλύψατε όλα τα ερωτήματα, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Νταμάτο είπε, έθεσε ένα ερώτημα προς τον κύριο Ζέγκερ, μήπως θέλετε να λάβετε το λόγο και να απαντήσετε στο θέμα αυτό εν συντομία. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα νομίζω ε, τέθηκαν σε μένα. Το πρώτο είχε να κάνει με την αξιολόγηση αυτή καθ' αυτή των ε, σχέσεων ε, εταιρική σχέση, ας πούμε. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, γεγονότα που για τα οποία ενημερωθήκαμε σύμφωνα με την, από την μελέτη μάλλον. Και βεβαίως είναι διαφορετικές οι καταστάσεις μεταξύ χωρών και εντός της ίδιας χώρας, μεταξύ των περιφερειών. Όλα εξαρτώνται από τον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας αλλά και άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει να μελετηθούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί εις βάθος για να ε, καταγράψουμε τις βέλτιστες πρακτικές και προτείνεται να προετοιμαστούν κάποια έγγραφα για τις περιφερειακές εταιρικέ σχέσεις ή να συμπεριληφθεί και το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο στην προετοιμασία, στη φάση της προετοιμασίας των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε την σωστή εμπλοκή όλων των επιπέδων της ε, διακυβέρνησης. Ε, βεβαίως υπάρχουν διαφορές και στην ποιότητα. Η τεχνική βοήθεια πολλές φορές ε, καλύπτει μόνο τα βασικά καθήκοντα και ε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες στα λεγόμενα νέα κρατημέλη. Η τεχνική λοιπόν επικούρηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προετοιμασία των εκτελεστικών αυτών ε, εγγράφων. Θα πρέπει να, ε, υπάρχει κυρίως στην προετοιμασία των ε, προγραμμάτων για να έχουμε και καλύτερη ποιότητα τελικά. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί βεβαίω που είναι διαθέσιμοι όπως η ανταλλαγή των πρακτικών αλλά και άλλα θέματα. Ωραία, ευχαριστώ. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Θα παρακολουθούμε φυσικά το θέμα. Αναφέρατε και μια ακόμη ανάλυση που θα παρουσιαστεί εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συμμετοχή σας. Κύριε Ζάγκαρ και σας, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στην ημερήσια διάταξη. Επόμενο σημείο, πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ε, έκθεση πρωτοβουλίας για, την ολοκληρωμένη, για τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχή 2014-2020 ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση και τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Η κυρία Τόμασιτς είναι η συγγετριά μας. Στην, ε, στην πολιτική συνοχή και στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ε, υπάρχουν δύο νέα εργαλεία για να επιτευχθούν οι στόχοι της εδαφικής συνοχής η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και η ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση. Η έκθεση πρωτοβουλίας έχει ως στόχο να αξιολογήσει αυτά τα, πρώτα, αυτά τα εργαλεία και να καταγράψει τα εμπόδια που υπάρχουν στην εφαρμογή τους. Σήμερα η, η συγγήτριά μας, η κυρία Τόμασιτς, θα αναφέρει τις βασικές, της αρχικές σκέψεις της για, την, ε, για το σχέδιο ε, έκθεσης που θα υποβάλει στις 3 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε τον Φλεβάρι του επόμενου έτους. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε 35 λεπτά μόλις για τη συζήτηση και να δώσουμε αμέσως το λόγο στην κυρία Τόμασιτς για την παρουσίασή της και μετά να συνεχίσουμε με την ε, συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. στο διάστημα 2014-2020 η Κομισιόν έχει θέσει την έμφαση στην εδαφική συνοχή. Οι δημοσιονομικές προοπτικές που περιλαμβάνονται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι φορά τα διαφορετικά ταμεία και των επενδύσεων λαμβάνουν υπόψη και αυτά τα εδαφικά μέσα όπως το CLLD και το ITI. Πρόκειται για εργαλεία για να ε, ε, συνοδεύσουν τις ε, άλλες δραστηριότητες. Θα πρέπει να βοηθήσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και την τοπική ανάπτυξη. Και υπάρχουν και κάποια όρια και υπάρχουν και προτεραιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να, για τον λόγο αυτό να υπάρξει ο απαραίτητο συντονισμός και την τήρηση νέων κανόνων που ακριβώς περιλαμβάνουν σε αυτό το νέο στρατηγικό πλαίσιο. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας έχει ως στόχο να αξιολογήσει τις πρώτες εμπειρίες και αποτελέσματα από πλευρά των μελών και τις βέλτιστες πρακτικές κατά τη στιγμή που θα εφαρμόσουν τα προαναφερθέντα μέσα. Και αυτό στο πλαίσιο της ε, γενικής εκτέλεσης της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης την περίοδο 2014-2020. Επίσης ε, θα αναλύσει και τον διάφορα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζει κατά την εφαρμογή του και να εξετάσει ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να εφαρμοστούν. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει διάφορε προκλήσει οικονομικέ και κοινωνικέ. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση περιφερειακή και εδαφική. Επίση απαιτείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ε, χαρακτηριστικά των επιμέρους ε, εδαφών. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πάμε πέρα από τα υφιστάμενα όρια. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια περαιτέρω δέσμευση των διαφόρων επιπέδων διαχείρισης για να υπάρξει ο απαραίτητο σύντονισμό σχετικά με την εκτέλεση αυτών των κοινών στόχων. Το άρθρο 7 προβλέπει 50% ε, των μέσων του Περιφερειακού Ταμείου σε αυτές τις ολοκληρωμένες ε, δράσεις περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης ε, προβλέπει και αυτή την ε, ολοκληρωμένη ταφική επένδυση. Αυτή η ITI, όπως λέγεται, η ολοκληρωμένη ταφική επένδυση, λαμβάνει υπόψη και επιμέρους προγράμματα για κάθε κράτος μέλος, λαμβάνει υπόψη τις χαρακτηριστικά κάθε μιας περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ε, η ε, πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD. Η δημόσια διοίκηση δυστυχώς δεν ε, τηρεί αυτές τις δεσμεύσεις και βλέπουμε να υπάρχει συχνά μια έλλειψη συνειδητοποίησης ε, και συνεργασίας ανάμεσα σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Έτσι απαιτείται να βρούμε μια στρατηγική η οποία θα ενημερώνει αλλά και θα επικεντρώνεται στις δράσεις ε, των δημοσίων αρχών χρειάζεται να ε, υπάρξουν ε, να υπάρξει ανάληψη ευθυνών για τον λόγο λοιπόν αυτό να απαιτούνται στρατηγικές αναπτυξιακές σταθερές μακροπρόθεσμες Απαιτείται λοιπόν η απαραίτητη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό. Απαιτείται χρόνος και μέσα προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι στρατηγικές και αυτή η πρωτοβουλία των κοινοτήτων. που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την εμπειρία των τοπικών αυτών αρχών. Όλα αυτά χρειάζονται 6, μήνες, 6 με 12 μήνες για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία όλος αυτό ο περίπλοκος μηχανισμός. Είναι περίπλοκος ο μηχανισμός διότι οι τοπικές αρχές είναι ήδη ε, περίπλοκε. Μπορούμε όμω ε, κατά τη διάρκεια αυτή τη προσπάθεια ε, να δούμε, βρούμε νέες ιδέες και έτσι ε, η νέα οδηγία αναφίβολα μπορεί να ε, οδηγήσει σε επιτυχία. Το πέραν των διαφορών που υφίστανται ανάμεσα τα διάφορα κράτη-μέλη, θα πρέπει να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα, π.χ. στην δυνατότητα των ε, τοπικών αρχών, των δαπάνε των νοικοκυριών, δημόσιες επενδύσεις, δημόσιες ταπάνες ένδια, κοινωνικός αποκλεισμός, κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να γίνουν, υπάρχουν ανταλλαγές πληροφοριών. Χρειάζονται επίσης μηχανισμοί παρακολούθησης και μηχανισμοί αξιολόγησης προκειμένου να απαντηθούν, να ανταποκριθούν πάνω στις ανάγκες των διαφόρων αρχών. Αυτό δεν είναι ζήτημα τυπικό απλά για να διολογήσουμε δαπάνες, αλλά θα πρέπει να κατορθώσουμε να υπάρχει μια ε, αποτελεσματική ενημέρωση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Χρειαζόμαστε επίσης κατάλληλα μέσα αξιολόγησης και παρακολούθησης. Πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και να προσαρμόσουμε την στρατηγική ανάλογα. Να, συνδέσουμε, να συνδυάσουμε στόχου σαφεί και μετρήσιμους μέσω μηχανισμών αξιολόγησης. Αυτό επιτρέπει στους, ε, να αναπτύξουμε πολιτικές πιο αξιόπιστες και πιο προσαρμόσιμες στις ανάγκες η διαδικασία επιλογής προγραμμάτων θα πρέπει να είναι διάφανη και να μην οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση. Χρειάζεται επίσης ένα σύστημα λήψης απόφασης που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων. Πρέπει να διαφωνιστούν όλες οι φάσεις σε αυτή την αλυσίδα. Παρομοίως πρέπει να εγγυηθούμε την ανάληψη των ευθυνών και υπάρχει και κάποιο όργανο προσφυγής. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια συστήματα διατησίας ε, αντικειμενικά αλλά και μέτρα συμφιλίωσης προκειμένου να ξεπερνάμε διάφορα προβλήματα διοικητικής ε, φύσης ή οικονομικής που ενδεχομένως να προκληθούν κατά διάρκεια διαφωνιών Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων χρειάζεται την ε, ανάγκη ύπαρξης των απαραίτητων οργανισμών για την ε, εφαρμογή της. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απλούστευσης πρέπει να έχουμε μια κοινή βάση για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Οι συστάσεις ε, σε μια χώρα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε μια άλλη χώρα αν δεν ληφθεί υπόψη το σύνολο. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς ε, θα μπορέσει να ε, αξιολογηθεί η ITT και η CLLD. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστώ τους ε, σκιώδες ηγητές για την συνεργασία τους και αυτή ήταν μια πρώτη μου έκθεση και σίγουρα θα, ε, θα ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε τώρα το λόγο αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Μπούδα, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια για την παρουσίασή της και για την ε, πολυθετική συζήτηση που κάναμε στο Στρασβούργο. Όλοι οι μηχανισμοί που μπορούν να δημιουργηθούν από την Κομισιόν με στόχο να διευκολυνθεί η περιφερειακή ανάπτυξη είναι φυσικά καλόδεκτοι. Είναι χρήσιμο να μιλάμε για αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό ανεργίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι μηχανισμοί και όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες θα πρέπει να τύχουν απλοποίηση των διαδικασιών τους. Πολύ συχνά συμφωνώ με εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών και όλοι τους διαμαρτύρονται για την υπερβολική ε, γραφειοκρατία η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να κάνει κάτι για τα θέματα αυτά. Πρέπει οι μηχανισμοί αυτοί να γίνουν πιο εύκαμπτοι, πιο ευέλικτοι. Πρέπει οι εμπλεκόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να καταλήξουν στις κατάλληλες λύσεις. Θα πρέπει να μπορούν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των περιοχών τους. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για την αρχή τη επικουρικότητα, ότι οι αποφάσει θα πρέπει να λαμβάνονται στο επίπεδο το οποίο είναι πιο κοντά στον πολίτη, στο τοπικό επίπεδο, γιατί το τοπικό επίπεδο είναι αυτό το οποίο γνωρίζει καλύτερα ποιε είναι οι ανάγκες και ποια είναι τα πρόσφορα εργαλεία για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει πολλά λοιπόν προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να είναι τμήμα τη έκθεση. Να δούμε επίση πώ θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη απόδοση για τις επενδύσεις που γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο πολλές φορές. Πολλές φορές οι δημοσιονομικές πολιτικές, η φορολογία η οποία συλλέγεται σε περιφερειακό επίπεδο πηγαίνει κατευθείαν στο κεντρικό θεσσαυροφυλάκιο ενό κράτου και η διανομή αυτών των ποσών σε περιφερειακό επίπεδο δεν είναι πάντα ισοδίκαια. Θα ήταν χρήσιμο όμως να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους φόρους που συλλέγονται σε περιφερειακό επίπεδο πάλι σε περιφερειακό επίπεδο χωρίς να εμπλέκεται το εθνικό επίπεδο. Θέλω, θα έρθω και πάλι σε επαφή με την κυρία Σιγήτα για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κυρία Ροντρίγες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Σιγήτρια για την ε, ε, έκθεσή και για το ανοιχτό πνεύμα σε διαλόγου που έχει δείξει. Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο είναι στεναρό και συνεκτικό και καταδεικνύει τη σημασία της πολιτικής συνοχής. Ο στόχος μας προφανώς στην Περιφερειακή Επιτροπή είναι να διευκολύνουμε τη χρήση των εργαλείων συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τα δύο αυτά εργαλεία τα οποία λειτουργούν σε εδαφικό επίπεδο και σε επίπεδο αστικού χώρου, το CLLD και το ITI <clears throat> και γνωρίζουμε επίσης ότι η εφαρμογή αυτών των δύο εργαλείων έχει σαν στόχο να επιτευχθούν και οι στόχοι της Ευρώπης 2020 και γι' αυτό το έργο μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας θα επιτρέψει να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη και που θα ενισχύσει την βιωσιμότητα και την αστική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις εδαφικές ανάγκες των περιφερειών πάντα σε ένα, πλε... σε ένα πνεύμα εθνικής συμφωνίας και συνένεσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε υπερπεριφερικές περιοχές, ιδίως αυτές οι οποίες είναι νησιωτικές. Είναι απαραίτητο εκεί να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τοπικών περιφερειακών παραγόντων και των εθνικών αρχών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο είναι φανερό ότι εκεί υπάρχουν οι ειδικέ γνώσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί περισσότερο βάρος στο τοπικό επίπεδο. Έχουμε μιλήσει σε μια προηγούμενη συνεδρίαση για την ανάγκη να υπάρχουν οι προϋπολογισμοί τεχνικής αρρωγής προς το τοπικό επίπεδο, αλλά φυσικά δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των δομών που δημιουργούνται. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια λογική αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας να επανακινητοποιήσουμε τις υπηρεσίες που υπάρχουν για να μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το εγχείρημα. Θα πρέπει να συμμετέχουν λοιπόν οι αρχές αυτές από την αρχή. Πιστεύω λοιπόν ότι μια τέτοια ευελιξία <clears throat> που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη μας συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει κατανοητή και να εφαρμοστεί και σε νομικό πλαίσιο που σημαίνει ότι όλοι οι παρεμβέντες στην σύλληψη, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση των προγραμμάτων λαμβάνουν υπόψη αυτή την παράμετρο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνονται με συμπερίληψη και της διάσταση της υπερπεριφερειακής κατά περίπτωση ή της νησιωτικής φύσης ορισμένων εδαφών. Και θα πρέπει να γίνει αυτή η εργασία σε επίπεδο συνεργασίας όλων των επιπέδων για να υπάρξει μια καλύτερη μορφή καθορισμού των πολιτικών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο είναι προφανές για μένα από τα έγγραφα τα οποία ανέγνωσα είναι ότι η πιο μεγάλη δυσκολία προκύπτει γιατί γιατί δεν γίνεται κατανοητός ο ρόλος που πρέπει να έχει το τοπικό επίπεδο στα έγγραφα αυτά. Υπάρχει, υπάρχει μια τάση να δημιουργούνται περισσότεροι φορείς για την επίλυση διαφορών και διαφωνιών. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις ε, ιδιαιτερότητες των ε, ορισμένων περιοχών που είναι υπερπεριφερειακές και είναι απαραίτητο να υπάρξει η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και η λογική των εργαλείων αυτών να γίνεται πάντα υπό το πρίσμα των προτεραιοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα ήταν χρήσιμη μια αξιολόγηση η οποία δεν θα έχει τυπικό χαρακτήρα για την εκτέλεση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να γίνεται με στόχο τη βελτίωση των βελτίστων πρακτικών σε ό,τι αφορά αυτά τα προγράμματα και την καλύτερη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω στους αδέλφους, ε, πρέπει να είναι σύντομοι. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων πάνω στο θέμα και προτού να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεμάτο να σας πω ότι ζήτησα από τον κύριο Πότζακ ε, να συνεχίσει με τη μέσα διάταξη διότι πρέπει να βγω να συναντήσω το μεσηκλημένο μας ε, τον ε, Ρωμάνο Υπουργό. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα περιοριστώ, στην, περιοριστώ στην ουσία και στις προτάσεις. Αυτά τα δύο μέσα δημιουργήθηκαν για να υπάρξει η διάδραση ανάμεσα στα διάφορα περιφερειακά περιφερειακές διοικήσεις. Όλοι θα ήθελα να μάθουμε πώς θα λειτουργήσουν και η τοπική ανάπτυξη συμμετοχικής ε, φύσης θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2017. Σημαντικές ε, προθέσεις και οι προσδοκίες, αλλά αυτά τα δύο μέσα κινδυνεύουν, εάν δεν συνοδεύονται από ανάλυση των ε, αναγκών των εδαφών, να ε, καταστούν ένα αυτεπίστροφο για τις τοπικές και περιφερειακές ε, διοικήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα απλούστευσης, κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και θα εξετάσουμε μάλλον αργότερα. Ε, τονίσω ότι στην γνωμοδότηση της επί των Περιφερειών αναφέρεται ότι καμία μεθοδολογία δεν χρησιμοποιήθηκε με τρόπο ξεκάθαρο για την εφαρμογή των ET και των CLLD. Θα ήταν λοιπόν επιθυμητό από πλευρά Κομισιόν μια ε, μεγαλύτερη ενημέρωση. Τέλος, η αρχή της εταιρικής σχέσης το είδαμε και σήμερα το πρωί είναι μια, ένας από τους βασικούς άξονες της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν ως εκ τούτου να εφαρμοστεί και ο ορισμός των στρατηγικών θα πρέπει να ε, μπλέκει και τους, ε, τις τοπικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Συγκήτρια. Θα ήθελα να αναφερθώ στα ίδια επιχειρήματα τα οποία ανέφερα και την πέσμα στο Στρασβούργο. Λέω να πω ότι αυτά τα μέσα ε, ιδρύθηκαν για την βελτίωση της γραφικής ε, ε, προσέγγισης και κινδυνεύουμε να μην πετύχουμε τις προσδοκίες μας λόγω της περιπλοκότητας του θέματος και όπως είπε η κυρία ε, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη ανάμεσα στους εθνικούς εταίρου και τους τοπικού εταίρου που μπορούν να ε, ζημιώσουν την επίτευξη του στόχου. Οι στόχοι, μάλλον εργαλεία είναι δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω της διαφορετικής ε, διοικητική δομής. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν πάντα τις απαραίτητες προφορίες σχετικά με το σχέδιο που θέλουν να υλοποιήσουν οι δημόσιες αρχές δεν είναι πάντα πρόθυμες να ζητήσουν ευρωπαϊκούς φόρους, ε, το, πόρους για την περαιτέρω απλούστευση, κάτι που είναι κατεπήγον. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να τηρήσουν οι περιφερειακές αρχές είναι πολύ περιοριστικά. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι αποθαρρύνει πολλούς από τους φορείς σχεδίων να ζητούν ε, χρηματοδότηση από την Ένωση. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το γεγονός ότι πολλές από τις τοπικές διοικήσεις δεν έχουν τις απαραίτητες δυνατότητες και γνώσεις για να υποβάλουν τους φακέλους της αρμόδιες αρχές και ε, πολλές φορές η κατάσταση αυτή αποθαρρύνει τις ε, τοπικές διοικήσεις από το να παρουσιάζουν φακέλους και όπως είπε ο προλαλής σας, υπάρχει συχνά επικάλυψη με άλλα εργαλεία. Στην Γαλλία υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία άλλοι επικαλύπτονται και θα πρέπει να κάνουμε το ισχύον σύστημα λίγο πιο απλό, να το αποστέψουμε με λίγα λόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω, μάλλον να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Γιάκοβιτς που είναι ε, σκιώδης ηγητής. Θα είμαι σύντομος. Το ITI και το CLLD δεν είναι, είναι καινούργια μεν μέσα, αλλά δεν είναι και τόσο πια καινούργια γιατί είχαμε το Leader Plus που ήταν ουσιαστικά ο προάγγελος του CLLD. Και επίσης είχαμε και προηγούμενες εκδοχές του ITI. Το ITI κυρίως για αστικές περιοχές προσφέρει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μπορεί κανείς να συνδυάσει και, ταμεία, και χρηματοδότηση από τον από το Κοινωνικό Ταμείο, από το Ταμείο Συνοχής, από την Περιφερειακή Ανάπτυξη για να ε, διεξάγει μια πολιτική ας πούμε για την ε, αγορά εργασίας. Οπότε ουσιαστικά μπορούσαμε να πειραματιστούμε με αυτά τα στοιχεία. Η Κομισιόν θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φιλόδοξη. Αν δείτε τι συστάσεις και αν δείτε την εμπειρία που έχει η Επιτροπή των Περιφερειών και διαβάσετε και τι εταιρικέ σχέσει, τις ε, συμφωνίε εταιρικών σχέσεων που υπάρχουν, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλέ περιφέρειε και χώρες που θέλουν να δουλέψουν πάνω στα CLD και τα ITI, αλλά που βλέπουν ότι υπάρχουν διοικητικοί φορείς στα κρατημέλη που δεν θέλουν να εκχωρήσουν οποιαδήποτε εξουσία στο τοπικό επίπεδο. Που σημαίνει ότι τα εργαλεία αυτά, τα μέσα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν, να εκτελεστούν επαρκώ. Ελπίζω λοιπόν ότι η κυρία Τόμασιτ και η έκθεσή τη θα αποτελέσει μια ενθάρρυνση, ένα έναυσμα για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία, να εφαρμοστούν σωστά και θα αποτελέσουν και ένα έναυσμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δει πού μπορεί να δοθεί υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη, γιατί κάποια κράτη-μέλη ε, ανησυχούν ιδιαίτερα και προβληματίζονται για τούτα τα εργαλεία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί θα έχουμε να ακούσουμε την κυρία Υπουργό Θα ήθελα να δώσω στο τέλος και το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία της κυρίας Τόμασιτς που είναι εισηγήτρια για το θέμα αυτό είναι καλόδεκτη. Νομίζω ότι η συνεργασία πρέπει να είναι μια συνεργασία ποιότητας. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία θα ευνοήσουν την εδαφική ανάπτυξη. Χάρη σε αυτά τα εργαλεία μπορούμε να πετύχουμε πολλά στην πολιτική συνοχή. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των κρατών μελών και όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εξ ονόματος των Πρασίνων. Θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε τα ET και τα CLLD. Διακόπτει ο πρόεδρος τον ομιλητή. Και 5% των ταμείων του Περιφερειακού Ταμείου έχουν προορισμό τα CLLD και τα ITI, κάτι το οποίο φυσικά είναι σημαντικό. Η κυρία Τόμασίτς έχει συνοψίσει πολύ σωστά τους στόχους αυτούς. Τώρα το θέμα είναι να δούμε ποια είναι τα εμπόδια για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό το οποίο δεν χρειάζεται να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες γραφειοκρατικές στρώσεις. Αντίθετα πρέπει να τις μειώσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία στην εφαρμογή αυτών των εργαλείων Επίσης πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη κατάρτιση του προσωπικού το οποίο θα λειτουργήσει και θα διαχειριστεί αυτά τα, εργασία, αυτά τα εργαλεία. Χρειάζεται επίσης να προσφύγουμε και σε εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Αυτό το τοπικό επίπεδο φυσικά έχει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης. Δεν αρκεί να δημιουργήσουμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να έχουν και του απαραίτητου μηχανισμού που θα του βοηθήσουν αυτά τα οποία δημιουργούν να είναι πιο επωφελή και αυτά που προτείνονται στην έκθεση τη κυρία Τόματσιτς είναι πράγματι προ τη σωστή κατεύθυνση. Ακολουθεί. Η κυρία Μπρέσολα Εφίε. Είμαι εγώ ίδιος. θα ήθελα να πω τα εξής για τα λεγόμενα της εισηγήτριας για το τι λειτουργεί και το τι δεν λειτουργεί στα CLD και τα EDI. Αυτό το οποίο προτείνεται είναι μια διαδικασία εκ των κάτω προς, τα άνω που αντανακλούν τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και οδηγούν σε μέτρα τα οποία συνάδουν με τις τοπικές ανάγκες. Αλλά η DG Regio εξακολουθεί να επιμένει λέγοντας ότι οι δραστηριότητες CLLD θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το περιεχόμενο των λειτουργικών προγραμμάτων και έτσι οι δραστηριότητες εκτός των προγραμμάτων αυτών δεν μπορούν να τύχουν υποστήριξης. Η εφαρμογή λοιπόν των προγραμμάτων, εάν εκφεύγει των λειτουργικών προγραμμάτων, δεν μπορεί να χρηματοδοτηρείται. Μα πιστεύουμε ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν την χρηματοδότηση προγραμμάτων και στρατηγικών που δεν είναι καθορισμένες εκ των προτέρων στα πρότυπα λειτουργικά προγράμματα. Αυτό είναι και το νόημα αυτών των στρατηγικών. Επομένω, οι στρατηγικές του CLLD θα πρέπει να εξυπηρετούν το γενικό στόχο των λειτουργικών προγραμμάτων, αλλά όχι του συγκεκριμένου στόχου του. Από ό,τι ξέρω, η DigiRegio ζητά κάτι το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Με το να έχουμε αποφάσει εκ των άνω προς τα κάτω δεν θα λειτουργήσουν τα πράγματα και αυτό έρχεται σε αντίφαση με τη σωστή μέθοδο για τα CLLD. Και τώρα δίνω το λόγο η κυρία Τόμασιτς για να κάνει τα συμπεράσματά της μετά από τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις σας και τις, για τις προτάσεις και τις συστάσεις σας. Το σχέδιο έκθεσης θα το εξετάσουμε στις 30 Νοεμβρίου ή 1 Δεκεμβρίου και φυσικά η έκθεση αυτή θα είναι έτοιμη για, για όλους σας σε δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο σε... στην κυρία Τζούντι Τρόσα που είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση Εμείς έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ε, δαφική συνοχή στην νέα προγραμματική περίοδο, θα το έχετε καταλάβει αυτό, και έχουμε εισαγάγει νέα εργαλεία όπως το ITI και το CLLD και το άρθρο 7 για την βιώσιμη ε, ανάπτυξη. Ε, πάντα είναι καλό να βλέπει κανείς τις εμπειρίες και να δει τι λειτουργεί και τι όχι επί τόπου Παρόλο που πρέπει να πω ότι ακόμα είναι πολύ νωρί. Οπότε όλα τα κράτη-μέλη και οι τοπικέ αρχέ και οι περιφερειές του προ το παρόν ε, προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτά τα νέα μέσα, προετοιμάζουν τις στρατηγικέ τους σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης να τονίσω ότι οι κανόνες είναι αρκετά ε, ευέλικτοι στο πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα εργαλεία κάτι που δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσει κανείς με απλό τρόπο αυτά τα μέσα, αλλά και με περίπλοκο ή πιο δύσκολο τρόπο αν το επιθυμεί. Συμφωνώ με πολλές από τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν ότι όντως υπάρχει ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και φυσικά πάντα μας ενδιαφέρει να ακούμε και συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτό το σκοπό. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δημιουργία δυνατοτήτων, και αυτό είναι ένα τομέα όπου χρειάζονται κοινέ προσπάθειε και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο τη Κομισιόν. Από την πλευρά τη Κομισιόν έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο, το δίκτυο αστική ανάπτυξη, που έχει στόχο να υποστηρίξει όλε τι αστικέ αρχέ που θα εφαρμόσουν τι στρατηγικέ του άρθρου 7. Υπάρχουν πολλέ προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε η προσέγγιση πολυ... η πολυταμιακή, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί επιτόπου. Υπάρχουν δυνατότητες για τα κράτη-μέλη να την ε, χρησιμοποιήσουν. Επίσης να πω ότι του χρόνου θα κάνουμε δύο μελέτες, μία για το άρθρο 7 και τη στρατηγική ITI, όπου θα δούμε το περιεχόμενο της στρατηγικής αυτής, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα από αυτές τις πρώτες εξελίξεις και επίσης θα γίνει μία μελέτη για το CLLD από κοινού με τις τέσσερις γενικές διευθύνσεις που εφαρμόζουν αυτό το εργαλείο. Οπότε ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του επόμενου έτους να έχουμε πιο συγκεκριμένα, πιο εις αποτελέσματα από αυτές τις δύο προσεγγίσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και τώρα περνούμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Σεβίλ Σαϊντέ, Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης α, της Ρουμανίας. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή μας έχει την πρακτική να καλεί υπουργούς από τα κράτη-μέλη για να μοιραστούν μαζί μας τις ε, εμπειρίες τους από την πολιτική συνοχή. Η Επιτροπή ΡΕΤΖΙ ήταν ένας ε, ενεργός συνομοθέτης από κοινού με το Συμβούλιο στα πλαίσια, για το νέο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η προσοχή μας λοιπόν τώρα στρέφεται στο πώς εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Γι' αυτό ε, έχω την χαρά ε, να ε, καλωσορίζω εδώ την κυρία Σάιντε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας για να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της από την πολιτική συνοχής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ε, επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων και στην εφαρμογή τους στα πλαίσια της, ε, του συντονισμού που παρέχει το Υπουργείο της. Θα ζητήσω από την ε, Υπουργό να κάνει μια σύντομη παρουσίαση, 15 λεπτών το πολύ, και μετά θα δώσω το ε, λόγο στα μέλη, ξεκινώντας από τους συντονιστές. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Να θέσετε ερωτήσεις εντός ενός λεπτού για να μπορούμε να είμαστε και ε, στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων μας. Φαντάζομαι ότι Ε, και οι σοσιαλιστές θα πάρουν το λόγο γιατί ήταν αυτοί που είχαν προτείνει την πρόσκληση αυτή προς την Υπουργό. Ε, βεβαίως θα συνεχίσουμε την πρακτική αυτή. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, μέλη του ε, Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιόν σας στο πλαίσιο αυτής της ε, έκτακτης ε, συνεδρίασης. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας και εκ μέρους της ε, ομάδας της οποία διευθύνω στο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ για την στήριξή σας, για τη σημασία του περιφερειακού προγράμματος και για την στήριξη των προγραμμάτων από την Ένωση στη Ρουμανία να πω ότι το μέτρο N 3 στην ε, Ρουμανία υπήρξε μια εξαιρετική βοήθεια, εξαιρετική στήριξη. Οι στόχοι που έχουμε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης είναι εξή. Επιθυμούμε η Ρουμανία να καταστεί μια επικράτεια ανταγωνιστική με συνοχή και πολύ καλά ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουμε ανταγωνιστικοί με τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι αστικές περιοχές αλλά και τα υπόλοιπα εδάφη. Να υπάρχουν λοιπόν συνοχή και να επιτρέψουμε σε όλους τους ε, κατοίκους ε, της χώρας ε, να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες αποτελεσματικές. Για το λόγο λοιπόν αυτό είναι ζωτική σημασία οι πολίτες και οι κοινότητες να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Πρέπει να έχουμε σχέδια που θα οδηγήσουν στην ευημερία και στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ως εκ τούτου, το βασικό μέλημα του Υπουργείου το οποίο ηγούμε είναι να τονίσουμε την κατάλληλη προσαρμογή των προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται σήμερα από τα, από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ω εκ τούτου, δεδομένου το επίπεδο ανάπτυξη τη Ρουμανία, χρειάστηκε να εφαρμόσουμε ένα μείγμα πολιτικής και μείγμα εργαλείων μέσων. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε μία μόνο εναλλακτική. Βασικό μας, βασική μας πρόκληση σήμερα και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι η βασική μας πρόκληση είναι η εγγύηση συμπληρωματικότητας ανάμεσα στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους και τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρέπει να εγγυηθούμε τη χρηματοδότηση των ε, τοπικών δομών. Προκειμένου τώρα για την χρηματοδότηση που προέρχεται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Σήμερα η Ρουμανία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της στην ε, περίοδο 2014-2020 και δεδομένου αυτού σε εθνικό επίπεδο λάβαμε όλα τα μέτρα που επιβάλλονταν προκειμένου να επιτρέψουμε την εφαρμογή και υλοποίηση αποτελεσματική των Διευθυντικών ταμείων. Επιθυμώ να κάνω αναφορά τώρα στα επιχειρησιακά προγραμμάτα 2007-2013. Ο συνολικό προπολογισμό είναι τη τάξη του 3,9 δις ευρώ. Σήμερα, που σα απευθύνω το λόγο, κατορθώσαμε να πετύχουμε ένα ποσοστό απορρόφηση τάξη του 63%. Κάτι που αντιπροσωπεύει τα ποσά τα οποία ε, πραγματικά ε, πλήρωσε, κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτήσαμε υποδομέ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μερικά παραδείγματα, πάνω από 2.000, ε, ε, χιλιόμετρα ε, δρόμων. όπω επίσης δημιουργήσαμε 29.000 θέσει εργασία με τη χρηματοδότηση σε μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίση για το 2014 2020 που αυτή τη φορά θα έχουν ένα προπολογισμό πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή 6,7 δις ευρώ, θα επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε 9 από τους 11 θεματικούς στόχους των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Θα ήθελα να αναφερθώ στην χρηματοδότηση των οδών που επιτρέπουν την σύνδεση με το δίκτυο TNT. Το θέμα της ε, ε, της ενίσχυσης ε, που χορηγούνται για, τις, ε, για τα σχολεία αλλά και για την κατασκευή ε, μονώσεων στα κτίρια. Θέλουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την καταχώρηση στο κτηματολόγιο πάνω από 5 εκατομμυρίων εκταρίων το μεγαλύτερο δίδαγμα που συναλλάγουμε από την τελευταία προγραμματική περίοδο 2013 και που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το 2014 είναι πως ε, απαιτείται να, ε, ε, να βελτιώσουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν συμμετείχα σε πολλές συνεδριάσεις με μέλη της Επιτροπής και επίσης διδαχτήκαμε από τα σφαλματά μας. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να υπογράψουμε τις συμβάσεις για όλους τους δικαιούχους σε μια περίοδο πολύ πιο σύντομη από αυτήν που καταγράφηκε κατά την προηγούμενη περίοδο. Επιθυμούμε οι δικαιούχοι των προγραμμάτων να μπορέσουν να τα εξελίξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην χρειαστεί να καταλήξουμε στο τέλος της περίοδου δίχως ε, να έχουμε μπορέσει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κεφάλαια. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα καλό σύστημα για την αποδέσμευση των πληρωμών όπως ε, πράξαμε από το 2014 διότι λειτουργήσε πολύ σωστά, πολύ καλά. Ε, διδαχθήκαμε λοιπόν από τα σφάλματα του παρελθόντος και εφαρμογή των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 να στεφθεί από επιτυχία. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω πως το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης έχει 12 προγράμματα συνεργασίας εδαφικής φύσης με ένα προπολογισμό 1,4 δις ευρώ. Ένα παράδειγμα να αναφέρω που είναι καλό παράδειγμα και δείχνει την επιτυχία της περιφερειακής συνεργασίας. Πρόκειται για τη συνεργασία ανάμεσα στη Ρουμανία και την Βουλγαρία. Το ποσοστό απορρόφησης αυτού του προγράμματος είναι της τάξης του 73%. Και μια που σας ανέφερα για τις ανάγκες εξασφάλισης της ειρηματικότητας ανάμεσα στα περιφερειακό πρόγραμμα και το εθνικό, θα σας πω ότι το μέσο που χρησιμοποιεί το Υπουργείο μας είναι το ε, πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε η ρουμανική κυβέρνηση, χρηματοδοτείται από τον κρατικό προπολογισμό και που στηρίζει την τοπική και περιφερειακή διοίκηση σε όλη την Ρουμανία. Επιπλέον, της χρηματοδότησης ε, σε περιφερειακό επίπεδο των το ε, περιφερικής, τοπικής, ανάπτυξης ε, αφορά συστήματα για την πρόθεση σχολικών κτηρίων και βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ σωστά συνδυαζόμενο με το άλλο πρόγραμμα το κοινοτικό. Ποιε είναι οι προσδοκίε μου από αυτήν την συνεργασία μαζί σα. Επιθυμώ να υπάρξει μια ανοιχτή εταιρική σχέση μαζί σα με τις υπηρεσίες ε, της Γενικής διεύθυνση Ρέτζο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διότι η Ρουμανία πρέπει να μπορέσει να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ε, κονδύλια που τη διατίθενται και οι πολιτικές ε, ανάπτυξης να προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της Ένωσης. Από πλευρά μου θεωρώ πως θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρξει μια ατζέντα ε, συναντήσεων όπως η σημερινή με όλους τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι συναντήσεις αυτές να διεξάγονται με τη συμμετοχή των ε, ε, της περιφερειακής διάθεση της Κομισιόν. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, διασφαλίσουμε την ευημερία των ε, πολιτών μας και των χωρών μας. Μπορώ να σας ε, πω ότι όλοι οι συνεργάτες μου είναι διαθέσιμοι για μια πιο στενή συνεργασία. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Μπορείτε ιδιαίτερη να βρεθώ σήμερα ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι το θεματολόγιο του Υπουργείου σας για τη διαχείριση των διαφορετικών πόρων είναι ακριβώς το ίδιο της Επιτροπής Περιφερειακών ε, Θεμάτων. Είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και συζητούμε εδώ και χαίρομαι που συμπίπτουν με τα δικά σας προβλήματα. Κυρίε και κύριοι, τώρα έχετε το λόγο. Θα είπαμε να ξεκινήσουμε με τους συντονιστές με την κυρία Κρέελ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας κυρία Υπουργέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ και μπορούμε να σας καλωσορίσουμε. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να συναντηθούμε στο Βουκουρέστι Δεν είναι εύκολο το έργο σας, φυσικά. Πρέπει να αντιμετωπίσετε ως υπουργό πολλά θέματα τα οποία είναι δύσκολα και πιστεύω ότι ήδη έχετε εξασφαλίσει να αυξήσετε το ποσοστό απορρόφησης στο 36% στο 63% συγγνώμη και αυτό δεν είναι φυσικά το 100% αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη αποτελεί μια επιτυχία από τη δική σας πλευρά. Είπε ήδη η Πρόεδρος μας ότι, ότι έχουμε φυσικά τα ίδια θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Επιτροπή μας όπως είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε και μια ακρόαση η οποία θα αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών στην πολιτική συνοχής και εγώ θα ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα να ακούσω από εσά πώς εσείς στη Ρουμανία έχετε οργανώσει τις διοικητικές διαδικασίες και πώς σκοπεύετε να τις απλοποιήσετε, να απλοποιήσετε και τα συστήματα πληρωμών. Αν μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και εμείς να ξέρουμε για τη δική μας εργασία πώς κινήσετε Ξέρουμε ότι και η Κομισιόν έχει δημιουργήσει μια υψηλού επίπεδο ομάδα για την απλοποίηση των διαδικασιών. Δεύτερο τώρα. Εγώ υποστηρίζω ιδιαίτερα αυτό που λέτε ότι θα πρέπει οι Υπουργοί Περιφερειακής Πολιτικής να συναντώνται σε τακτικά διαστήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διεκδικεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολύ καιρό να υπάρξει ένα, ένα Συμβούλιο Υπουργών Περιφερειακής Πολιτικής και Συνοχής. Αυτό δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Ίσως όμως στην επόμενη Προεδρία θα μπορέσουμε να δώσουμε και μια όθηση περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Ελπίζω στο μέλλον να μπορέσει να γίνει δυνατό αυτό, γιατί φυσικά οι Υπουργοί Περιφερειακών Θεμάτων και Συνοχής έχουν σημαντικές ευθύνες. Επίσης, ένα τρίτο σημείο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαιρετήσει το σχέδιο Juncker για τις επενδύσεις. Θα ήθελα να ξέρω αν εσείς θα μπορούσατε να μας πείτε πώς τα μέσα αυτά τα οποία θα έρθουν στην διάθεσή μας, στη διάθεση των περιφερειών, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με τα ήδη υπάρχοντα διαφορετικά ταμεία για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ, Λίπρόδος. Ο κύριος Γιάκοβ Τσίτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Μιχαήλοβα, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την Υπουργό για το γεγονός ότι δέχτη την, ε, πρόθεση, την ε, πρόσκλησή μας και έχει έρθει ως τις Βρυξέλλες για να συναντηθεί μαζί μας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας να γνωρίσουμε καλύτερα ποιες είναι οι σκέψεις της κυρίας Υπουργού και πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στα κράτη-μέλη η παρουσίασή σας ήταν πάρα πολύ σημαντική για όλους μας και την παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή. Ήθελα τώρα να κάνω ένα ερώτημα προς ε, εμάς που θα μπορούσαν να κάνουν φυσικά βουλευτές και από άλλες χώρες και κυρίως από τις ε, χώρες που έχουν προσχωρήσει πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η άποψη που έχετε για το πρόβλημα της απορρόφησης των πόρων. Είναι ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να είναι επίκαιρο σε πολλές χώρες. Εγώ ήμουνα κυβερνήτης της Ίστρια, μιας περιφέρειας στην Κροατία και διαπίστωσα ότι ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζεται εκεί είναι η έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με το βαθμό αποκέντρωσης ή μη αποκέντρωσης ενός κράτους. Έχει να κάνει με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να έχουν οι περιφέρειες ενός κράτους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως το οποίο μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην απορρόφηση των κονδυλίων και να την εμποδίσει. Η Κροατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά θα χρειαστεί να επενδύσουν πολύ περισσότερες επενδύσεις, ιδιαίτερα <clears throat> για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και οι πόλεις και οι περιφέρειες ξέρουν πολύ καλά πού και πώς και σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Εγώ προσωπικά έχω εμπειρία στα θέματα αυτά εδώ και 5, 6, 7 ακόμα χρόνια όμως βλέπω ότι η συγκέντρωση, η συγκεντρωτική διοίκηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι περιφέρειες στη Ρουμανία έχουν επαρκή χρηματοδοτική ικανότητα για να μπορούν με τα δικά τους εργαλεία να λειτουργήσουν και να εκμεταλλευτούν αυτά που δίνονται από την Ευρώπη στην πολιτική συνοχή. Σε ευχαριστώ, Λίκη Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Μια απλή ερώτηση, αλλά πρακτικής φύσης. Αν υπήρξαν δυσκολίες και κάποια παραδείγματα ενδεχομένως να μας δώσετε, αναφορικά με τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσατε στη διαχείριση των πόρων, εφόσον η χώρα σας έχει εισέλθει εδώ και λίγο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Madame la Ministre. Vous avez... Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Αναφερθήκατε σε... στην έλλειψη απλούστευσης. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα, διότι αναφέρατε ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τα σφάλματά μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί την περίοδο 2014-2020. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε την κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω από ίδια εμπειρία ότι δεν είναι εύκολο να περάσει κανείς από το ένα σύστημα στο άλλο. Είναι όντως δύσκολο να γίνει αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε πού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μεταξύ της συνεργασίας του κράτους, των περιφερειών και, των, και του τοπικού επίπεδου. Αν βρήκατε λύση, πώς εξελίχθηκε, τι προτείνατε και σε άλλες ε, χώρες που έχουν απαλλαγή από το κομμουνιστικό σύστημα για να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από δυόμιση χρόνια περίπου ή τρία χρόνια, είχαμε μία αντιπροσωπεία η οποία πήγε στην Ρουμανία στην Τιμισοάρα και στα σύνορα στο Δούναβι Ρουμανίας-Βουλγαρίας και εκεί αυτό που είδαμε και ακούσαμε ήταν ότι υπήρχαν παράπονα για το θέμα της αποκέντρωσης και της περιφερειοποίησης και επίσης της μεταφοράς των ευθυνών προς τις ε, περιφέρειες της Ρουμανίας γιατί υπήρχαν προτάσεις ε, για προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο και για τη διεξαγωγή αυτών. Ε, τα παράπονα ήταν ότι δεν είχαν προχωρήσει λοιπόν όλα αυτά και γι' αυτό ρωτώ. Η διαρθρωτική πολιτική είναι περιφερειακή πολιτική. Κυρίως Βεβαίω, όταν ε, μεγάλα, τα, τα μεγάλα κράτη αποδίδουν τι ευθύνε στι περιφέρειέ του για να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα. Υπήρχε τότε στην ε, ρουμανική κυβέρνηση ε, μια πρόταση νόμου για την ε, περιφερειοποίηση και την αποκέντρωση της διοίκησης. Πόσο έχει προχωρήσει αυτή, οι περιφέρειες τώρα σε αυτή τη νέα περίοδο, την προγραμματική, θα έχουν περισσότερη επιρροή στην διάρθρωση των, των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που ασχολούνται ακριβώς με την εφαρμογή όσων αποφασίζουμε εμείς εδώ σε ε, πολιτικό επίπεδο. Ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν για την εφαρμογή. Μιλήσατε για 63% ανάληψης απορρόφησης των κονδυλίων. Τι ε, βοήθεια χρειάζεστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό απορρόφησης. Επίσης, ως πράσινη, η ε, στόχη του κλίματος και η επίτευξή τους με ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε ότι έχουμε επενδύσεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, έχετε μιλήσει πάρα πολύ για τη δημιουργία, για την κατασκευή δρόμων, έχουν υπάρξει σκέψεις για το πώς θα γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές, ας πούμε οι επενδύσεις στους σιδηροδρόμους. Μιλήσατε για την ενεργειακή απόδοση. Αυτό το σκέφτεστε στα πλαίσια των μεταφορών. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ψηφίζουμε πάνω σε μια έκθεση σήμερα για τις, περιφερ, για τις κοινότητες και πώς αυτές μπορούν να ενταχθούν στις πολιτικές συνοχής. Η Ρουμανία έχει μια μεγάλη μειονότητα Ρωμά και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες. Τι κάνετε για να τις συμπεριλάβετε και να τις κάνετε να εποφεληθούν από αυτά τα περιφερειακά κονδύλια ή άλλα ταμεία στη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Πότζακ έχει το λόγο για την επόμενη ερώτηση. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ το ίδιο ερώτημα είχα να θέσω με τον ε, κύριο Τσέλερ. Πώς ε, οι τοπικές ε, και οι περιφερειακές αρχές μπλέκονται στην όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων Και θα ήθελα να θέσω κι άλλο ένα ερώτημα. Στην Τσεχία και εμείς έχουμε κάποια προβλήματα όταν μιλούμε για θέματα απορρόψης κονδυλίων. Η ποσόσταση μέχρι το 2013 ε, ήταν 26,5 δισεκατομμύρια. Από αυτά θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε μόλις 2,5, δηλαδή περίπου 10% του κατρεμημένου ποσού. Εσείς ξέρετε σε ποιο βαθμό θα είσαστε έτοιμοι να απορροφήσετε τα κονδύλια αυτά. Έχετε κάποιο στοιχείο για το τελικό ποσοστό. Ευχαριστώ. Κύριο Σάριμον, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όποιος ε, γνωρίζει την ε, πραγματικότητα και το παρελθόν μπορεί να αντλήσει διδάγματα για το μέλλον. Όταν έχουμε την έκθεση του 2014 για τα οικονομικά συμφέροντα, η Ρουμανία είχε 52 περιπτώσεις απατών και ατασταλιών στην πολιτική ε, περιφερειακό και 133 σε επίπεδα τελειών και τασταλαιών. Αυτά είναι ένας μεγάλος αριθμός σε σχέση με άλλα κράτη. Υπάρχει κάποιο σχέδιο από τη δική σα πλευρά για το 2015 να, έχουν, να υπάρχουν λιγότερες ατασταλίε και λιγότερες περιπτώσει απάτη στο μέλλον. Ευχαριστώ και το τελευταίο ερώτημα από τον κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το, την κυρία Υπουργό που ήρθε ε, σήμερα ενώπιόν μας. Ένα σύντομο ερώτημα για σας σε σχέση για το θέμα της διοικητικής αποκέντρωσης στη Ρουμανία. Η περιφερειοποίηση στην ε, ε, Ρουμανία σε διοικητικό επίπεδο θα μπορούσε να δίνει σε υψηλότερο επίπεδο ε, απορρόφησης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και αυτοί εμποδίζουν την απορρόφηση των πόρων. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας σκέφτεται λοιπόν να προχωρήσει σε μια αποκέντρωση των διοικητικών ε, αρμοδιοτήτων για να βελτιωθούν τα ποσοστά απορρόφησης. Σας ευχαριστώ Λεκύη Πρόεδρος. Κλείσαμε με τις ερωτήσεις, με τον πρώτη, την πρώτη ομάδα ερωτήσεων. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για να δώσετε απαντήσεις στα πολύ ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα. Βλέπετε ότι έχουμε πραγματικά τα ίδια θέματα που μας απασχολούν όπως και εσάς τους Υπουργούς Περιφερειακών Θεμάτων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Είναι γεγονός πως ε, οι ερωτήσει αυτές ε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και οι απαντήσεις που θα δώσω θα αφορούν πολλές ερωτήσεις ε, τώρα σχετικά με την απλούστευση. Να σας πω ποια είναι τα βασικά μέτρα τα οποία λάβαμε για αυτή την περίοδο προγραμματισμού σε σχέση με την προηγούμενη. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την επιλογή των προγραμμάτων, έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα της εφικτότητας των προγραμμάτων. Ένα πρόγραμμα μπορεί να γνωρίσει διάφορες φάσεις. Αρχικά υπάρχει η μελέτη, η αρχική, η οποία καθορίζει την αξία της επένδυσης. Μετά η μελέτη που αξιολογεί την ε, σημασία του έργου και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και όλα αυτά τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της περίοδου 2007-2013 είχαν ως αποτέλεσμα να απαιτείται 1,5 έως 2 χρόνια προτού να εγκριθεί το πρόγραμμα. Δηλαδή από τη στιγμή που το το πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία υπογραφής προγράμματος 24 μήνες χρειάζονταν να παρέλθουν. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτή η διάρκεια της περίοδου έχει μειωθεί, η φροντίζουμε να τη μειώσουμε τώρα από 24 σε 4 μήνες και κάτι ακόμα. πάνω στο οποίο θέλουμε να μειωθεί η περίοδος. Θέλουμε να υπάρξει ένας, ένας οδηγός προς τους δικαιούχους. Μιλάμε για την επαλήθευση επιτοπίως των όσων αναφέρει ο δικαιούχος στο πρόγραμμά του το οποίο έχει καταθέσει και όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται με την παρουσία του ενδυνάμει δικαιούχου της χρηματοδότησης. Επιθυμούμε λοιπόν να μην απαιτείται πάνω από ένα μήνας, 30 μέρε για την αξιολόγηση όλων αυτών των ζητημάτων. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μία σύμβαση χρηματοδότηση στάνταρ. Είτε πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση κάποιων οδών ή την ανακαίνιση σχολείου. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ε, έχει υιοθετήσει και ένα νέο νόμο αναφορικά με τις ε, δημόσιες αγορές. το πιο, το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προ, προ, περίοδου η νομοθεσία σχετικά με τις αγορές ε, του δημοσίου δημιουργούσε διάφορες δυσκολίες. Τώρα έχουμε μια νέα νομοθεσία η οποία απλούστευσε ουσιαστικά την όλη διαδικασία, την κατέστησε πιο διάφανη και πιο γρήγορη. Ένα άλλο μέτρο και επιτρέψτε μου τώρα να ε, συγχωνεύσω ερωτήσεις σε μία απάντηση Μιλάμε για τους μηχανισμούς ε, καταβολής των πληρωμών. Όταν έφτασα το 2012 στο Υπουργείο, ήμουν υφυπουργό και το πρόγραμμα για την περίοδο 2011-2013 είχε μια απορρόφηση της τάξης του 12%. Μετά από ένα χρόνο κατόρθωσα η ομάδα μου και εγώ να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό απορρόφησης σε 45-50%. Πώς κατέστη δυνατόν αυτό. Το δικό μας ποσοστό απορρόφησης ήταν τόσο χαμηλό λόγω του μηχανισμού επεξεργασίας των ετοιμάτων επιστροφών στους δικαιούχους. 80% των δικαιούχων αυτού του προγράμματος ήταν δημόσιες αρχές δημαρχία, σχολιά, νοσοκομεία. Φυσικά οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζουν πολύ καλά το μηχανισμό αυτόν τον οποίο έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να λάβει, να χρηματοδότηση ως δικαιούχος χρειάζεται πρώτα να καταβάλεις το ποσό και να αποδείξεις ότι η δαπάνη όντως πραγματοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει πως εγώ ως δικαιούχος πληρώνω ένα τιμολόγιο προς τον κατασκευαστή και έπειτα αποστέλω το τιμολόγιο στην αρχή, διαχειριστική αρχή η οποία με τη σειρά της την αποστέλει στην DG Regio και ζητάει την επιστροφή του δαπάνης λοιπόν λόγω του συστήματος αυτού χρειαζόμασταν μεταξύ 6 και 8 μήνε μήνες για να μπορέσει ο δικαιούχος να λάβει τα χρήματα το οποίο είχε δαπανίσει. Γι' αυτό λοιπόν κατορθώσαμε να εφαρμόσουμε έναν άλλο μηχανισμό. Ξοφλήσαμε τη τιμολόγια με κονδύλια του, από τον Εθνικό Προπολογισμό. Δημιούργησαμε λοιπόν ένα ταμείο για να επιστρέψουμε στους δικαιούχους τα χρήματα τα οποία είχαν ήδη δαπανίσει. Και χάρη σε αυτό το ταμείο που δημιουργήσαμε και χάρη στο ταμείο αυτό οι δικαιούχοι μπορούσαν να καταβάλουν τα, τα έξοδα του έργου. ο οποίος διόχος απευθυνόταν σε αυτό το ταμείο το οποίο είχαμε συσταθεί. Εδώ λοιπόν οι λύσεις που μπορέσαμε να εφαρμόσουμε οι οποίες ε, στέθησαν από επιτυχία και χρησιμοποιήθηκαν όμως και για άλλα προγράμματα στη Ρουμανία και αυτό το μέτρο θα συνεχιστεί και την περίοδο 2014-2020. Μου θέσατε και κάποια άλλα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την αποκέντρωση, την περιφερειοποίηση, τι συμβαίνει στη Ρουμανία. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, ως επικεφαλής Υπουργείο εφάρμοσε, μάλλον, ε, ε, δημιούργησε την απαραίτητη νομοθεσία διότι η περιφερειοποίηση είναι μια διαδικασία που αποβαίνει προς όφελος της κοινωνίας. Αλλά για να κατορθώσουμε να την εφαρμόσουμε στην πράξη για να αποκτήσει νομικό, νομικό πρόσωπο οι περιφέρειες ε, της Ρουμανίας έπρεπε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Αυτή η τροποποίηση του Συντάγματος είναι αντικείμενο συζητήσεων στο Κοινοβουλίο μας. Και γνωρίζουμε ότι δεν είναι μια πολύ απλή διαδικασία αυτή απαιτείται χρόνος, διότι μετά από την εξέλιξη από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να οργανώσουμε και ένα δημοψήφισμα του αντίον κατορθώσαμε να πετύχουμε τα εξή. Υπάρχει μια, μια, διοικητική, μια διαχειριστική αρχή. Έχουμε οκτώ στατιστικές περιφέρειες που ασχολούνται με την περιφερειακή ανάπτυξη. Εκεί συμμετέχουν ε, δημαρχία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και αυτό το Συμβούλιο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι το αρμόδιο για την κατάρτιση της στρατηγικής ε, που καθορίζει τις προτεραιότητες αυτής της περιφέρειας. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης στηρίχθηκε σε αυτές τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης. Και μολονότι η διαχείριση ε, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, οι αποφάσεις και ο καθορισμός των αναγκών καθορίζεται από τους δικαιούχους και από τις περιφερειακές αρχές. Το πρόγραμμα, το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker ε, ευχαριστώ για την πρωτοβουλία αυτή. Το Υπουργείο μας, όπως και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα Υπουργεία, εργάστηκαν προκειμένου να εντοπίσουν τα καλύτερα προγράμματα που θα μπορούσαν να αυξήσουν το επίπεδο ανάπτυξη τη ε, χώρα μα. Και πάντως ένα άλλο ερώτημα. Φυσικά ε, και έχουμε ανάγκη από περισσότερου πόρου από όσους λαμβάνουμε σήμερα από τα ευχησιακά προγράμματα. Το πρόγραμμα Juncker είναι μία λύση. Μπορούμε να καλύψουμε λοιπόν όλες τις ε, ανάγκες μας ε, σε ρηφά τη χρηματοδότηση διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Juncker και να πάρουμε χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε άλλα προγράμματα. Δηλαδή με λίγα λόγια, τι εννοώ. Αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού που είχε αποδοθεί στα προγράμματα αυτά μπορεί να αναδιανεμηθεί προς τις τοπικές περιφερειακές αρχές προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές τους. Που βεβαίως δεν είναι τόσο σημαντικά όσο αυτά τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσω του προγράμματος Juncker. Θα χαρώ πολύ αν αυτές οι συναντήσεις με τους άλλους υπουργούς ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης θα μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα. Ακόμα και σε άτομο επίπεδο θα χαιρόμουν πάρα πολύ να συζητώ μαζί σας, να έχουμε σε επαφή με την DG ε, Regio, την υπηρεσία της Κομισιόν, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι θετικά. Εγώ έχω μια εμπειρία διοικητική 25 ετών και παραπάνω και 15 χρόνια συν σε ό,τι αφορά χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκού φορεί. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε από εμά, μεταξύ των υπουργών, μεταξύ των συναδέλφων, κερδίζει με το να εργάζεται μόνος του, να εργάζεται σε ένα κενό αέρος. Πρέπει να είμαστε σε επαφή, να κάνουμε αυτέ τι συναντήσει ώστε να μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι τι επιτυχίε μα τις εμπειρίες μας, θετικές ή αντικές, να συζητήσουμε για τα θέματα της συμπληρωματικότητας, για την ανάγκη να έχουμε απλοποίηση των διαδικασιών. Στα προγράμματα πληρωμών παγκοσχάρη επιτύχαμε μια απλοποίηση, η οποία ήταν μια πολύ επιτυχής εμπειρία. Να μπορέσουμε λοιπόν από κοινού να βελτιώσουμε τα ποσοστά απορρόφησης των κονδυλίων και με την υποστήριξή σας και με την υποστήριξη των συναδέλφων από την DG Regio μπορούμε να βελτιώσουμε όλες τις διαδικασίες αυτές. Τους οδηγούς, τα εγχειρίδια, τα εγκόλπια, όλα αυτά τα οποία απεικονίζουν τα μέτρα που έχουμε θεσπίσει, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς ως μέλη του Κοινοβουλίου να μπορείτε να είστε επιπισμένοι ότι η Ρουμανία και άλλες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορθό και διάφανο τρόπο και επανέρχομαι στο θέμα του αν έχουμε ένα γενικό σχέδιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε <clears throat> τις ατασταλίες και τα θέματα ενδεχομένων απατών κτλ. Υπάρχει μια απόφαση της κυβέρνησής μας, ένα διάταγμα το οποίο ρυθμίζει όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ατασταλίες επί τη βάση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιαδήποτε μορφή ε, ενεργειών που είναι κολάσιμες θα την χάνει κυρώσεων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα χρηματοδοτούμενα σχέδια και προγράμματα. Δεν ήταν εύκολο να το πετύχουμε αυτό. Παραδείγματος χάρη. Έχουμε ένα σύστημα δημοσίων διαγωνισμών και προμηθειών που διαπιστώσαμε ότι δεν ευθυγραμμιζόταν με όλες τις ε, ε, προδιαγραφές και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφαση λοιπόν που λαμβάνετε τώρα, έχουμε αλλάξει το σύστημα αυτό και οι δικαιούχοι μας, για πολλούς από τους δικαιούχους μας, αυτή η αλλαγή ήταν πολύ δύσκολο να τη δεχτούν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ελπίζαν ότι θα μπορέσουν να τύχουν ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη εξανεμίστηκαν οι προοπτικές χρηματοδότησης. Κάποιοι άρχισαν να χάνουν ένα σημαντικό μέρος χρηματοδότησης που, στην οποία προσέβλεπαν 20% ή περισσότερο. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το περάσαμε για να ενισχύσουμε την εφαρμογή των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά λοιπόν προγράμματα, στο κεντρικό επίπεδο έχετε το Υπουργείο, αλλά μετά έχετε και τις τοπικές αρχές και ίσως οι τοπικές αρχές θα μπορούν τώρα να έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες να εκμεταλλεύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε αυτήν την αρχή δημοσίων διαγωνισμών σε κεντρικό επίπεδο που είναι αρμόδια για να αναλύσει τις προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν για τις δημόσιες προμήθειες, δημόσιους διαγωνισμούς και θα ελέγχουν όλες αυτές τις αιτήσει. Όταν παρουσιάζονται προβλήματα ή ε, συνθήκες οι οποίες είναι οι ατασταλίες θα υπάρχει μια διόρθωση κατά 25% και αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε δικαιούχος θα πρέπει να περάσει και πάλι από όλες τις αρμόδιες αρχές και μετά να καταθέσει πάλι η έκθεση. Έτσι η ρουμανική κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει τους δικαιούχους με το να παρέχει πόρους εφόσον οι ελεκτικοί μηχανισμοί έχουν δώσει το καλό σέχιν σε όλα τα επίπεδα και εφόσον έχουν εισαχθεί όλες οι απαραίτητες διορθώσεις, αυτό πρέπει να γίνει γιατί η προηγούμενη μας νομοθεσία δεν ήταν πραγματικά προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές. Αυτά κάνουμε λοιπόν για να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές. Και για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Φέραμε σε πέρας μια έρευνα με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δημιουργήσαμε ένα χάρτη όλων αυτών των κοινοτήτων που βρίσκονται στο περιθώριο. Λέμε ότι αυτό είναι ο χάρτης της ένδυας στη Ρουμανία, έτσι τον ονομάζουμε και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε πού βρίσκονται αυτές οι περιθωριοποιημένες κοινότητες σε επίπεδο περιφέρειας, γειτονιάς, ακόμα και δρόμου, να δούμε πού βρίσκονται αυτές οι κοινότητε με τα λειτουργικά προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε ήδη την διάσταση του CLLD, της τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητος και με τα προγράμματα της κυβέρνησής μας έχουμε ιδιαίτερα προγράμματα για να ευνοήσουμε τη στέγαση αυτών των περιθωρικοποιημένων κοινοτήτων. Και αυτό θα περιλάβει και την κοινότητα των Ρωμά μέσα στα περιφερειακά λοιπόν λειτουργικά προγράμματα, μέσα στα κυβερνητικά μας προγράμματα, δεν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε την κοινότητα των Ρωμά χωριστά από τις άλλες περιθωριακές κοινότητες. Θέλαμε να, να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση που σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις κοινότητες έχετε κάποιους Ρουμάνους αλλά έχετε και κάποιους Ρώμα. Δεν θέλαμε να έχουμε μια χωριστή προσέγγιση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά τα οποία έχουμε περάσει και έχουμε ενσωματώσει στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα θα βοηθήσουν όλες τις κοινότητες οι οποίες έχουν προβλήματα και βρίσκονται σε περιθωριακή κατάσταση. Να δω μήπως έχω ξεχάσει κάτι, κάποια άλλη ερώτηση ή όχι. Uh, am avut Α, ναι. Υπήρξε άλλη μια ερώτηση για την σύνδεση μεταξύ των κεντρικών και των τοπικών αρχών σε σχέση με τη βελτίωση του βαθμού απορρόφησης. Προσπάθησα να απαντήσω σε αυτό. Είπα ήδη ότι η κεντρική αρχή, οι κεντρικές αρχές ε, είναι αυτές οι οποίες στα πλαίσια του Υπουργείου για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη έχουν δημιουργηθεί αλλά δεν έχουν λόγο όταν μιλούμε για θέματα που άπτονται του περιφερειακού επίπεδου. Αμέσω δηλαδή σε τέτοιε περιπτώσει πηγαίνει η ευθύνη στι περιφερειακέ και τι τοπικέ αρχέ. Κανένα δεν θα πει λοιπόν στι περιφερειακέ αρχέ τι πρέπει να κάνουν και πώ να χρησιμοποιήσουν τα περιφερειακά κονδύλια. Βεβαίω υπάρχουν θεματικοί στόχοι πάνω στου οποίου βασίζονται και τα περιφερειακά προγράμματα. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι ανάγκε τη τοπική κοινωνία στη Ρουμανία. Ελπίζω τώρα να έχω απαντήσει σε όλε σα τι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Θυμόμαστε τα σχόλιά σας για, τους, για τις τακτικές συναντήσεις με τους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε βεβαίως αυτή την παράδοση. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τη συμμετοχή σας και καλή τύχη στο έργο σας στη Ρουμανία. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας ξανασυναντήσουμε όταν σε λίγα χρόνια θα μπορέσετε να μας πείτε πόσο υπέροχα προχωρούν τα πράγματα με την πολιτική συνοχή στη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους των μελών της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Okay, dear ladies and gentlemen, we continue. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε ψηφοφορία. Έχετε παρακαλώ τις ε, κάρτες σας ψηφοφορίας. Είναι έτοιμες για να τις χρησιμοποιήσετε. Thank you. Thank um, we vote today. Λοιπόν, ψηφίζουμε την έκθεση πολιτικής συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες. Ο κανονισμός, η νομοθεσία για την πολιτική συνοχή παρέχει οικονομική ενίσχυση για τις περιθωριοποιημένες περιοχές ε, στην Ήπεθρο για την ε, κοινωνική ένταξη, γιατί αυτό εμπίπτει στο πρόγραμμα στήριξης του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η περιφερειακή προσέγγιση για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 προσφέρει νέε ευκαιρίε για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τη ολοκληρωμένη ε, ε, εδαφική επένδυση και των ε, τοπικών πρωτοβουλίων που έχουν στόχο, πρωτοβουλειών που έχουν στόχο τι περιφερειοποιημένε κοινότητε. Η κυρία Ρέντκε, η συγκεντριά μα, παρουσίασε το σχέδιο εκθεσή τη το Μάρτιο του τρέχοντο με προθεσμία για γιατροπολογίας 2 ε, Ιουλίου. Είχαμε 214 τροπολογίες. Υπευλήθησαν εγκαίρως, εμπρόθεσμα και έχουμε και γνωμοδοτήσεις από άλλες δύο επιτροπές του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή Γυναικών. Η συγγήτρια επίσης προτείνει έναν αριθμό συμβαστικών τροπολογιών. Θέλετε να πάρετε το λόγο για πάρα πολύ λίγο, κύριε Ρέντκε, ή να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Να πω απλώς ότι ευχαριστώ τους συναδέλφους, Πρόεδρε, για τη συνεργασία τους και ελπίζω η έκθεση αυτή να καλύψει τα, όλα τα αιτήματα όλων όσων τους αφορά. Κυρία Κρέλ, κυρία Πρόεδρε, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά στην ημερήσια διάταξη έλεγε ότι θα ξεκινήσουμε στις 11.40 με την ψηφοφορία και τα μέλη μου δεν έχουν έρθει ακόμα. Παρακαλώ μπορούμε να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διαλυματάκι για να πάρω και τηλέφωνο του συναδέλφου γιατί θα ήθελα να είναι παρόντες οι συνάδελφοι στην ψηφοφορία. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Ε, συγγνώμη, σας, ε, το τρέχω πολύ το πρόγραμμα σήμερα. Ε, αλήθεια είναι ότι είχαμε πει 11.40 για την ψηφοφορία, οπότε Εντάξει, να κάνουμε ένα διαλυματάκι για να τα πούμε για ένα πεντάλεπτο. Ladies uh, Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είμαστε όλοι εδώ πλέον. Είναι όλα τα μέλη. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Είναι σημαντικό να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Οπότε ξεκινούμε με την ψηφοφορία για την έκθεση πολιτικής συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες. Η συγγήτρια η κυρία Ξεκινούμε με τη συμβαστική πρόταση 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 2. Παρακαλώ, κυρία εισηγήτρια, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, γιατί υπάρχει ένα λάθος ε, στον κατάλογο ψηφοφοριών. Εδώ βλέπετε στο δεύτερο κομμάτι λέει ιδιαίτερα η κατάσταση και στο τέλος, στην ε, σελίδα 18, λέει including, όχι in particular, για να είμαστε, έχει διορθωθεί ήδη δηλαδή στη σελίδα 18, είναι απλώς τεχνικό το λάθος για να είναι σαφές. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι θα ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Ευχαριστώ που μας το διευκρινίσατε. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Συμβαστική πρόταση, ε, δύο πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο ε, τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβιβαστική τρία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε, παρακαλώ να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής πρότασης 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Did you vote? The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Πάμε στη συμβαστική πρόταση 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 98. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε βεβαίως. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 98. Άρχιτη η ψηφοφορία της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. The vote Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην συμβιβαστική πρόταση 9. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 112, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 11, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ γιατί δεν βλέπω τα χέρια σας. Συμβαστική πρόταση 11. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. The vote is closed. Πέρας Εγκρίνεται. Παρακαλώ, σηκώνετε τα χέρια σας λίγο πιο ευκρινώς. Ε, συμβαστική πρόταση 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 185 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 185. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην συμβαστική πρόταση 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27. Όχι, ναι. Υπέρ, 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Έχει κάνει αντίρρηση? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ? κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 206, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 206, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 207. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 208. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε καλύτερα και αυτό. Ψηφίζουμε την τροπολογία 208 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Νομίζω απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε χρονικά την τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 8. Άρχιτη ψηφοφορία. Δεν άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 24 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 62, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 63, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στις συστάσεις της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Πάμε στην πρόταση α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Όχι. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Δι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τέσσερα υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε αυτό καλύτερα. Ψηφίζουμε λοιπόν το νούμερο 4, πρόταση του Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε. Ναι. 6. Σύσταση 6. Η 5 καταπίπτει. Σύσταση 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σύσταση 9. Υπέρ κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τη σύσταση 9 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. vote Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Σύσταση 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σύσταση 11. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύσταση 12. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14 και 15 καταπίπτουν. 16. Σύσταση 16. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 καταπίπτει, σύσταση 18, ψήφι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύσταση 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Σύσταση 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Σύσταση 21. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Ψηφίζουμε στις 22. Ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφορία. Έληξε. απορρίφθηκε. Σύσταση 23. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 ψήφι Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 25. Άρχιτη ψηφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Σύσταση 26. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα περνάμε στις τάσεις της Επιτροπής ε, Δικαιωμένων Ανθρωπών και Ισότητας του Φίλου. Σύσταση A. Ψήφι πέρ Κατά. Εποχές. Νομίζω πως εγκρίθηκε, αλλά ας επαληθεύσουμε καλού κακού. Ψηφίζουμε τη σύσταση A της Επιτροπής Γυναικών. Πέρα της ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. Σύσταση B. Ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σύσταση C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. E, υπέρ. Κατά αποχές ας επαληθεύσουμε σύσταση ή ε ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία Πέρασα. εγκρίνεται σύσταση F ψήφι πέρ κατά αποχές δεκτή G υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. H υπέρ κατά αποχές δεκτή. I υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. G υπέρ κατά αποχές δεκτή. K υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμόν 1, σύσταση υπαριθμόν 1. Όχι, κατα, καταπίπτει υπαριθμόν 1, καταπίπτει, περνάμε έτσι στην υπαριθμόν 2, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Υπαριθμόν 3, υπέρ. Κατά, αποχές, θα ελέγξουμε Σύσταση υπαριθμών 3. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας. Ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Συγγνώμη για αυτό το άσκηση που σας έβαλε να κάνετε. Σύσταση 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται οι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμόν 6 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε. Υπαριθμόν 6 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή υπαριθμόν 7 ψήφι υπέρ κατά εποχές δεκτή Υπαριθμόν 8 καταπίπτει Υπαριθμόν 9 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται Υπαριθμόν 10 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται Υπαριθμόν 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παριθμόν 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμό 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Υπαριθμό 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμό 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Υπαριθμό 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρθμο 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρθμο 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρθμο 19 υπέρ. Συγγνωμή, 20 γιατί δεν κάνει καλά Ψήφι υπέρ της 20 κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρθμο 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 καταπίπτει 24 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 συγγνώμη 26 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικός ε, άρχιδη ψηφοφορία. The Έληξε η ψηφοφορία. Έγινε δεκτή έκθεση. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ. Αποχωρήσατε τις αιθούσεις ησύχως και ταχαίως.